Meine Damen und Herren, und συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κατόπιν αιτήματος της διάσκεψης των Προέδρων πρέπει να σας ανακοινώσω κάτι. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου παρακαλεί να γίνει μια διόρθωση σε σχέση με τη σύσταση του Κοινοβουλίου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη Συμφωνία Σύνδεσης και τις Διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής ένωση Αζερβαϊτζάν σε μια ψηφοφορία έγιναν δύο τυπικά ε, σφάλματα γιατί κατατέθηκε μια προφορική τροπολογία χωρίς να συμφωνήσει η πολιτική ομάδα και η Προεδρεύουσα δεν ε, το συνειδητοποίησε και δεν ρώτησε αν 40 περισσότεροι βουλευτές ήταν κατά της τροπολογίας και αν θέλουν να εγερθούν. Αυτά είναι δύο τυπικά σφάλματα που σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τη διάσκεψη των Προέδρων επηρεάζουν ε, και ακυρώνουν μάλιστα την απόφαση και παρακαλώ να γραφεί στα πρακτικά ότι θα διαγραφεί αυτή η τροπολογία από την έκθεση για να επανέλθει η συνέχεια και οι συνέπειε αποφάσει του Κοινοβουλίου. Διαφωνείτε με αυτό. Όχι, ούτω λοιπόν και αποφασίζεται. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίε, θα ήθελα σύντομα να σας κάνω μια άλλη ανακοίνωση και να σας παρακαλέσω να συμφωνήσετε τα τελευταία χρόνια είχαμε πάντα μεγάλες συζητήσεις για τη συνεργασία των πολιτικών κομμάτων στην Αλβανία. Ήταν μεγάλη δυσκολία πάντα για να δοθεί καθεστώς υποψήφιας χώρες στην Αλβανία. Το Νοέμβριο άρχισαν διαπραγματεύσει μεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Μόλις συζήτησα με την ε, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αλβανίας και από ό,τι φαίνεται και μετά από παρέμβαση του ΟΑΣΕ στα μέσα Μαΐου θα έχουν καταλήξει σε μια κοινή θέση. Το συζητήσαμε και έτσι κι αλλιώς στις 14 Μαΐου θα έρθει εδώ και καλό θα ήταν κυβέρνηση και αντιπολίτευση από κοινού ε, να είναι σε θέση να παρουσιάσουν αυτό το αποτέλεσμα εδώ μαζί στην Επιτροπή μας. Εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον συζητάμε αυτό το θέμα και προσπαθούμε ως Επιτροπή να φέρουμε τα δύο κόμματα κοντά το ένα στον άλλο και καλό θα ήταν μια που θα συνεδριάζει και η Επιτροπή μας τότε να τους προσκαλέσουμε. Συμφωνείτε να στείλουμε αυτή την πρόσκληση. Να θέλουμε όμως και τις δύο πλευρές, έτσι, να έρθουν εδώ και τα δύο κόμματα να παρουσιάσουν τη συμφωνία τους. Ευχαριστώ πολύ και προχωρούμε. Ερχόμαστε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Σίβιτς ζητεί το λόγο. Σίβιτς προφέρεται έτσι. Ναι. Επό ότι η ψηφοφορία για την ε, ΑΚΑ ακυρώθηκε ε, για το Ισραήλ. Για ποιο λόγο, πώς την αιτιολογείται αυτή. Έχουμε μια γνωμάτευση της νομικής επιτροπής μας Τη νομική υπηρεσία, συγγνώμη, που είπε ότι υπάρχουν αμφιβολίες στην ερμηνεία της συμφωνίας. Και ε, αυτό θα μπορούσε να λυθεί με μια μονομερή διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Φιούλε, αρμόδιος επιτροπός, ε, διακήρυξε την περασμένη εβδομάδα ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια τέτοια δήλωση αλλά επειδή είχαν προβλήματα συντονισμού με τον ε, αρμόδιο επίτροπο εμπορίου και τα λοιπά, δεν πρόλαβαν να γνωμοδοτήσουν. Και το συζήτησα και με την κυρία Ντεκεζέρ και είπαμε να περιμένουμε για να βεβαιωθούμε ότι θα συνάδει και με ε, τα όσα έχουμε ζητήσει και ίσως γνωρίζετε. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες μέχρι να έρθει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην επόμενη ή μεθεπόμενη συνεδρίαση μα μπορούμε να αποφασίσουμε. Νομίζω ότι θα είχε νόημα κάτι τέτοιο και μπορούμε να οργανώσουμε και μια σταθερή πλειοψηφία ε, στην ε, Επιτροπή μας. Κύριε Σίβιτ, ευχαριστώ πολύ. Καλύτερο να υπάρχει μια πιο ισχυρή θέση. Είχαμε πολλούς δισταγμούς, κάναμε και πολλές συζητήσεις. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι θα περιμένουμε δηλαδή λίγες μέρες, ούτως ώστε... Πέστε μας μάλλον ε, πόσο καιρό θα περιμένουμε, ε, μέρες ή μήνες. Ε, και στην Ίντα τη θέση μας. Να τους πούμε τι, άποψη έχουμε εμείς. Ας περιμένουμε όμως το έγγραφο λοιπόν της Κομισιόν για να είμαστε σίγουροι. So, point nine. Mr. Baletskis. Το σημείο, ναι. Κύριε Παλέτσκης, έχετε να πείτε τίποτα ή τα πάτε όλα χτες. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Änderungsantrag Nummer 1. Ε, τροπολογία παριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές Υπέρ παρακαλώ τις τρία. Κατά. Νομίζω ότι απορρίφτεται, αλλά μάλλον να το ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 23-24. Aber dafür, dass der Herr Κύριος πήγε στο Λουξεμβούργο 4,5 ώρα το πρωί, επομένως είναι μεγάλη τιμωρία γι' αυτό. Ε, τέσσερα 4 κατά αποχές εγκρίνεται. 6 ε, είπε, κατά Νομίζω την ίδια πλειοψηφία και απορρίπτεται. Τσεκ. Η κυρία Βαϊντέρε θέλει να το ελέγξουμε. Πήρε και δεύτερη κάρτα και είναι έτοιμη να ψηφίσει δύο φορές. Πέρες ψηφοφορίες. Α, ένας όμως έχασε την κάρτα του. Τι έγινε, χάσαμε έναν. Λοιπόν, συμβαστική 1. Ε, ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, συμβαστική 2. υπέ. Ε, Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 3. Υπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία των 10 υπέ. Κατά αποχές συγκρίνεται. Η 14 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 15 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 είπε, κατά αποχές συγκρίνεται. 19 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 20 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 είπε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 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 4 σε δύο τμήματα χωρίς την εταιρική σχέση και συνεργασία υπέρ κατά ε, τώρα με την εταιρική σχέση και συνεργασία υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται επίσης. 31 31 υπέρ κατά όχι Α, όχι, όχι, ούτε και αυτή. Έχει καταπέσει. 33 πάμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τριάντα τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τριάντα πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική υπάρχει μόνο έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η προφορική του κυρίου Λανσμπέργης. Υπέρ. Κατά. Ξανά ρωτάω. Ψήφι υπέρ. Τη προφορική τροπολογία είναι του κύριου Λαντσμπέργης. Όλοι είναι υπέρ της αύξησης των αξιών μας. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. 42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 44 υπέρ. Υπέρ. 44. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τελική για το σύνολο της νομοδότησης, όπως τροποποιήθηκε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Με 48 ψήφους υπέρ και δύο εποχές. Συγχαρητήρια. Now we come to the report. Και τώρα ερχόμαστε στην έκθεση της κυρίας Βαϊτέρε. Έχετε να πείτε τίποτα, κυρία Βαϊτέρε. Ε, τελευταία σας επιθυμία. Potatoes with uh, <laughs> scrambled eggs. Amendment number 25, ε, ε, τροπολογία ψηφί Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. συμβασμός PA. Τι είναι το PA? A τον διορθώνουν τον πρόεδρο. Δεν το γράφουν καλά, πώς να το καταλάβω. Καλά είναι. Thanks. Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε. Σύμβα Α. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται στήρεται το πρόεδρος. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Όχι. 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μόνο το τμήμα για το άρθρο 7.2 ψηφίζεται. Υπέρ για αυτό το τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 11. Μόνο το τμήμα που αφορά το άρθρο 9.1 ψηφίζουμε. Υπέρ. Όχι, δεν είναι σωστό. Καταπίπτει γιατί το 48 ψηφίστηκε. That's Δεύτηκα, λέει ο πρόεδρος. Αυτό το άρθρο 9.1 μπορεί να... Το τμήμα για το άρθρο 9.1 μπορεί να ψηφιστεί. Α, όχι, διορθώνει ο πρόεδρος, το 9-2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και μετά έχουμε το 9-3, το τμήμα για το 9-3. Α, χάνει η κυρία Γκόμε, γιατί το δικό μου 9, 1, 2 και 3 περνάνε. Εγκρίνεται λοιπόν για το 11, 52. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 53, μαζί με την προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αποχή. The vote is closed. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, 23 κατά. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Απορρίπτεται, διορθώνει ο πρόεδρος. 18. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Υιοθετείτε. Πρώτη τροπολογία. Μαζί με την προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 20. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 4. Μαζί με την προφορική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. 5. Μαζί με την προφορική τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε μαζί, on block, τα παραρτήματα. Από την 56 μέχρι την 78. Συμφωνείτε? Υπέρ κατά, άποχες, σκληρή αλλά σαφής η απόφαση. Τώρα ψηφίζουμε την τροποποιηθήσα ε, γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότησης. Όπως τροποποιήθηκε λοιπόν, με ηλεκτρονικό τρόπο παρακαλώ. της ψυχοφορίας. Εγκρίνεται με 47 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια. No, we have to vote. Τώρα ψηφίζουμε την έκθεση της Σάρα Λάτφορντ. Είναι εδώ. Όχι. Ζητά συγγνώμη. Αλλά δεν θα μπορέσει να παραστεί σήμερα. Και την εκπροσωπώ. Αλλά δεν έχω τίποτα να πω. that you speak in the name of Sarah... Μιλάτε εν ονόματι της Σάρα. και δεν θα είχατε τίποτα. But, uh, send us all... Και άρα δεν έχετε τίποτα να πείτε. Ε, της ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Και ψηφίζουμε. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Μπορούμε να ψηφίσουμε on block. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. The vote is closed. Πέρας προφορίας. Τι λέτε. 19 υπέρ 32 κατά. Προφορική τροπολογία 1. Α, πρώτο τμήμα και δεύτερο τμήμα. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ και 22 ψήφους κατά και μία αποχή. Υπέρ του πρώτου τμήματο. Του δεύτερου του διορθώνει ο Πρόεδρος. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι κατά, λέει ο Πρόεδρος Ελληνιστή. The vote is 16 υπέρ, 32 κατά. Να το ξανατσεκάρουμε, Του ψηφιρίζουν από δίπλα. 38 και 48. Ε, δεύτερο block vote. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Υιοθετείτε. 42 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σημείο 5, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 5 βέβαια. Σε τέσσερα τμήματα. Μάλλον είναι σημαντική αυτή η τροπολογία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Ε, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή η τροπολογία. Πέρας πληροφορίες. 28 υπέρ, 23 κατά. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Κρίμα που η δική μου η ομάδα δεν με πιστεύετε. Ξέχασα να ψηφίσω. Πέρας ψηφοφορίας. Ω! Γκρίνεται λοιπόν. Σημείο τεσ... ε, τμήμα 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, άποχες, υιοθετείται. 7 υπέρ, κατά, άποχες, υιοθετείται. 8 υπέρ, κατά, άποχες, υιοθετείτε. 11 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Να τσεκάρουμε αν ψηφίσαμε. Τι έγινε με την 24. 22. Ψηφίζουμε. Κατά. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Υπέρ του 4. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Την 4. Εγώ νομίζω ότι εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. Πέρες ψηφοφορίες, 28 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άποχες, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Ε,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 Ο πρόεδρος λέει με 42 υπέρ, δύο ψήφους κατά, είναι λάθος, είναι 46. Yeah. Έχω πρόβλημα. Μερικοί από εμά δεν καταλάβαμε πάρα πολύ καλά τι ψηφίσαμε. Τι είπατε στην αρχή, ότι ακυρώθηκε, λέτε, η ψηφοφορία, αυτό που είχε αποφασίσει το κοινοβούλιο. Δεν κατάλαβα καλά. Μια ανακοίνωση που μας κάνατε στην αρχή. Έγινε μια προφορική τροπολογία δική σας, αν δεν απατώμε. Έτσι λέτε. Έτσι μου είπαν. Εγώ ήμουν απόν στην ψηφοφορία τότε στην Ολομέλεια. Αλλά η διάσκεψη των Προέδρων το επαλήθευσε και είπε ότι έγινε προφορική τροπολογία, όχι πολιτικής ομάδας, μεμονωμένη και στην... Ολομέλεια, μόνο οι πολιτικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν ε, τροπολογίες. Ένα αυτό. Δεύτερον, η Προεδρεύουσα εκείνη τη στιγμή δεν ε, ρώτησε αν διαφωνεί κανείς να ηγερθεί 45 προκειμένου. Σηκώθηκαν λέει ο κύριος Λατσπέργης, αλλά δεν ήταν αρκετοί. Ε, δεν το έκανε πριν την ψηφοφορία. Ε, το έκανε πολύ αργά. Δεν μπορέσαμε να το αποτρέψουμε γιατί ο ναι, κανονισμός δεν εφαρμόζεται ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε η ψηφοφορία με δύο τεχνικά σφάλματα και για το λόγο αυτό ακυρώνεται. Αυτό τι σημαίνει, Έλμαρ. Έχουμε πολίτμπυρό εδώ και είναι υπέρ της ε, κατοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ αυτό το πολίτμπυρό. Μα τι σχέση έχει αυτό με την ουσία, με τον τύπο έχει σχέση, με τον κανονισμό. Έχουμε ένα κανονισμό και είτε μας αρέσει η απόφαση είτε όχι, θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Μα ήταν σαφές το λέει ο κύριος Λατσπέργης σηκώθηκαν μερικοί, πολύ λίγοι, όχι αρκετοί εν περιπτώσει, αλλά εμένα μου είπαν, λέει ο πρόεδρος και συμφώνησε, ότι ε, αφορά και την δική μας επιτροπή και τη θέση της επιτροπής μας και αυτό οι φιλελεύθεροι, ο κύριος Φερχόφστα το απέρριψαν Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Ε, έχουμε έναν κανονισμό, είτε τον εφαρμόζουμε είτε δεν τον εφαρμόζουμε. Τον εφαρμόζουμε είτε μα αρέσει είτε δεν μα αρέσει. Όλοι όσοι ήταν στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα είδαν ότι αυτή η τροπολογία έχει βρει υποστήριξη. Αυτά που είχε προτείνει δηλαδή ο κ. Λανσπέργκης. anyway, has, Κοιτάξτε, πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες. Αν εφαρμόσουμε τους κανόνες, τι θα τους παρακάμψουμε δηλαδή. Ε, αντίθετα, ε, δρούμε εντελώς ε, διαφορετικά το Πολιτμπυρό. Ε, σεβόμαστε τους κανόνες. Οι κανόνες υπάρχουν για να μας προστατεύσουν. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε κανόνες με πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ε, ξεφορτωθήκαμε αυτή την απαράδεκτη τροπολογία. Οι δύο εκθέσεις δεν θα ήταν ε, συμβατέ. Θα ήταν αντιφατικέ ε, μεταξύ του. Δηλαδή, θα έστελνε δύο διαφορετικά μηνύματα εντελώ αντιφατικά και θα ήταν γελίο το κοινοβούλιο. Ε, η ομάδα μου, αν είχε καταλάβει περί τίνο επρόκειτο, θα είχε σηκωθεί. Αλλά δεν μα ειδοποίησαν. Ε, φαντάζομαι το Έλκετ την είχε υποστηρίξει την υπόθεση. Νόμιζα μάλλον, αλλά δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε κύριε Λασβέξ, έχετε αυτή την ε, απαράδεκτη συνήθεια να ρίχνετε, να εμφανίζετε ευνηδίω τέτοιε προφορικέ τροπολογίε τελευταία στιγμή. Δεν, είχα, δεν φέραμε αντίρρηση, αλλά αν είχαμε καταλάβει πριν ω πρόκειται, θα είχαμε φέρει α, αντίρρηση. Α, θα, δεν θα ήταν 14, θα ήταν 100 τόσοι, εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα είχε ανατραπεί και δεν θα είχε περάσει πραγματικά με όλου του κανόνε και με όλου του τύπου. Μην ανησυχείτε. Τέτοιε προφορικές τροπολογίες στην πολιτική δεν έχουν νόημα. Ήταν σαφέστατη προφορική τροπολογία για την αποχώρηση στρατευμάτων από κατεχόμενα εδάφη, όχι μόνο από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αν την είχατε διαβάσει, την είχατε καταλάβει. Ε, δεν έπρεπε να κοιμάστε. Και εγώ θα βάλω τέτοιες προφορικές τροπολογίες στην επόμενη έκθεση. Τι νομίζετε. Και αν κοιμάστε, να μην είστε στο κοινοβούλιο. Δεν θέλω να γίνει πολιτική συζήτηση, λέει η κυρία Βάιντερε. Αλλά αν υποστηρίζει το Κοινοβούλιο κάποια πρόταση, δεν νομίζω ότι το Προεδρείο έχει το δικαίωμα να την ακυρώνει. Θα πρέπει ε, αυτό το θέμα να ξαναπάει ενώπιον του Κοινοβουλίου για να αλλάξει. Δεν μπορεί το Προεδρείο τώρα να ακυρώνει αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Δεν είναι σωστή διαδικασία είναι εναντίον όλων των κανόνων. Είναι πολύ κακό προηγούμενο, έχω να πω. Δεν έχετε το λόγο όμως. Δεν είναι θέμα ουσίας, επαναλαμβάνω, είναι θέμα κανόνων. Τύπου, έχουμε ένα κανονισμό και οφείλουμε να τον εφαρμόζουμε. Και κάποιος το επαλήθευσε. Εγώ δεν το έκανα, ήμουν απόν κιόλα στην ψηφοφορία στο Στρασβούργο και δεν έχω άποψη γι' αυτό. Το θέμα δεν έχει νόημα ή δεν έχει νόημα. Έχουμε ένα κανονισμό, τον εφαρμόζουμε και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν έχετε εσείς απόδειξη ότι είναι λάθος η θέση, γράψτε στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι σέβομαι απολύτως τον συνάδελφο για την προσωπική του διαδρομή Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι σε αυτό το κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να είμαστε ένα κοινοβούλιο γράφει κρατικό. Ο καθένα θα πρέπει να έχει τα δικά του δικαιώματα. Και τώρα θα ήθελα να πω δύο πράγματα σε σχέση με την προφορική τροπολογία του συναδέλφου Λανσπέργη. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την ουσία. Αυτή η τροπολογία Εν πάση περιπτώσει, αυτή η παράγραφος στις δύο εκθέσεις ήταν αποτέλεσμα επιμελούς εργασίας και πολιτικής συνένεσης που αντικατοπτριζόταν και στις δύο εκθέσεις, και για την Αρμενία και για το Αζερβαϊτζάν. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Λανσμπέργκης δεν είχε την υποστήριξη του ΕΛΚ, δεν υπολογίσε αυτή την υποστήριξη να την καταθέση. Και δεν θα πω ότι εμείς ε, ε, εφησυχάσαμε όταν προσέστηκε, αλλά το λέω αυτό προς ε, σεβασμό προς τον κύριο Λασμέργης. Εγώ, για σεβασμό λοιπόν, δεν ζήτησα στους συναδέλφους του ΕΛΚ να σηκωθούν για να μπλοκαριστεί αυτή η τροπολογία. Τώρα, όσον αφορά, αυτά ήταν για το, την ουσία. πεις τώρα, πρέπει να πω ότι την τελευταία στιγμή παρουσιάστηκε η τροπολογία. Δεν υπήρχε στο κείμενο, δεν υπήρχε στον κατάλογο των προφορικών και υπήρξε λάθος εκ μέρους ε, του προεδρεύοντος εκείνη τη στιγμή. Διότι πρώτα απ' όλα δεν έθεσε το ερώτημα στην Ολομέλεια και δεύτερον όταν κάποιοι ε, εξέφραζαν την αντίθεσή του ε, δημιουργήθηκε η κατάσταση που δημιούργηκε και 40 και 14 ήταν κατά. Ήταν λοιπόν αυτή η διαδικασία πάρα, είχε δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Δεν έγιναν τα πράγματα σύμφωνα με την διαδικασία και δεύτερον, όντως 40 μέλη ήταν αντίθετοι. Πρέπει να πω λοιπόν ότι σωστή ήταν η απόφαση της, ε, του Προεδρίου, δεδομένου ότι κατέστρεφε την ισορροπία αυτή η τροπολογία της ισορροπίας της συνένεσης που είχε επιτευχθεί και άρα όταν δεν μπορεί, ε, δεν ακολουθείται η σωστή διαδικασία, αυτό μπορεί να συμβεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος uh, um, Δεν έχω να προσθέσω κάποια πράγματα. Πρέπει να πω όμως ότι οι σοσιαλιστές είχαν την ε, θέση η οποία διαμορφώθηκε συζήτηση. Δηλαδή, είχαμε την ίδια διατύπωση είχαμε αποφασίσει και στις δύο εκθέσεις. Και δεδομένου ότι δημιουργήθηκε σύγχυση με τον τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε η τροπολογία και δέθηκε θέμα με την διαδικασία, πρέπει να πω ότι εμεί, εγώ τουλάχιστον, δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί. πιστεύομαι, εγώ τουλάχιστον ότι περισκόθηκαν περισσότερο από 40 και δεν έπρεπε να ψηφιστεί. Τελικά καταλήξαμε στο αποτέλεσμα καταλήξαμε. Και χαίρομαι διότι η διάσκεψη των Προέδρων διευθέτησε το θέμα και έλαβε την απάντηση που έλαβε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν, λέει ο κύριος Τάνοκ, και ε, χαίρομαι που δεν πέρασε ε, λόγω τεχνικών προβλημάτων, αλλά ήταν και πρόβλημα διατύπωση. At first έλεγε στα αγγλικά, που δεν είναι σωστό. Έλεγε first ή immediately, δεν ξέρω τι. Ε, όχι at first, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι χρονική σειρά απαραίτητο πρώτα το ένα μετά το άλλο. Όχι αμέσως ασμένο, ξέρω εγώ. Ήταν και κακά αγγλικά, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν μεγαλύτερη η σύγχυση. Ε, διότι ε, γράφουν τροπολογίε κάποιοι που δεν είναι αγγλόφωνοι και η διατύπωση στα αγγλικά που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Λαντσπέργη δεν ήταν εύστοχη. Αυτό που ήθελε να πει να ζητήσει άμεση απόσυρση όλων των στρατευμάτων και από τον Αγκόνο Καραμπάχ και από τις γύρω περιοχές. Εννοούσε first, όχι at first, προφανώς ήταν σαφές. Και έχει νόημα κατά την πολιτική του άποψη, τη δική του. Ο κύριος Χάουιτ. Τα λέτε, Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να συζητούμε τώρα το περιεχόμενο, αλλά μόνο, μόνο τους κανόνες και τη διαδικασία. Έγινε αναγγελία της διαδικασίας και θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η κυρία Βάιτερε, δηλαδή, που είπε, ότι το θέμα αυτό ερωτά είναι σωστό η διάσκεψη των Προέδρων να είναι αντίθετοι και να απορρίψουν μία πρόταση που ελήφθη από την ε, Ολομέλεια. Θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό και πάλι ίσως ο Προεδρεύων εκείνη τη στιγμή διαπράξει κάποιο σφάλμα, Αλλά δεν ξέρω εάν ε, μπορούμε να δούμε τι ακριβώς είναι η σταπρωτικά. Πολύ σωστά έθεσε η κυρία Βάιταρη το ερώτημά της. Οποιαδήποτε λοιπόν αναφορά ε, στο στην ουσία τη απόφαση είναι άλλο θέμα. Και όπω ζήτησε θα πρέπει να ελέγξουμε στο πρακτικό να τι ακριβώς έγινε εκείνη τη στιγμή. Υποστηρίζω αυτό που Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιατεμάκη έχει τώρα το λόγο, η συγγήτρια. Arvoisa puhemies, kysymys on aivan selkeä menettelytapavirhe. Προφανώς είναι αυτή η έκθεσή μου και προφανώς υπήρξε σαφέστατο διαδικαστικό σφάλμα στην Ολομέλεια. Η, η ομάδα μου πιστεύει ότι σηκώθηκαν 40 άτομα στην αίθουσα της Ολομέλειας και όσοι καθόταν από πίσω, πίσω-πίσω και βλέπαν ας πούμε όλη την αίθουσα επιβεβαιώνουν ότι πάνω από 40 ήταν όρθιοι. Πάνω από 40 ευρωβουλευτές. Αμέσως μετά τη σύνοδο Ήρθα σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές για να τους πω ότι σηκώθηκαν πάνω από 40 ευρωβουλευτές και μάλιστα το συζήτησα και με μερικούς από εδώ. Πέρα από την ουσία, εγώ τώρα ασχολούμαι με τη διαδικασία. Προφανώς υπήρξε ένα διαδικαστικό λάθος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο μάλιστα διαδικαστικά λάθη έγινε. Α, κύριε Λανσπέργης τελευταίος, μετά θα τα πω εγώ όμως. Πρώτον, ο αρμόδιος να πει ε, πόσοι βουλευτές εγέρθησαν είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της ε, ε, Συνόδου, ο οποίος βλέπει μπροστά όλο τον κόσμο, δεν έχει μάτια στην πλάτη. Και είπε λοιπόν η πρόεδρος ότι ήταν λιγότεροι από 40. Μπορεί να υπάρχουν γνώμες ότι ενδεχομένω να ήταν και παραπάνω. Αυτά είναι κολοκυθιά. Ε, αυτό το πρώτο, at first. Μετά, χαίρομαι πάρα πολύ που κανείς δεν ε, συζητάει και δεν αφισβητεί το περιεχόμενο της τροπολογίας. Μόνο διαδικαστικά πράγματα συζητούμε τώρα. Σας ευχαριστώ που υποστηρίζετε το περιεχόμενο με τι άλλο. President, I am with the Κύριος Κασουλίδης, έχω την αίσθηση ότι οι τροπολογίες στην Ολομέλεια κατατίθενται εξ ονόματος μιας πολιτικής ομάδας, με την έγκριση της πολιτικής ομάδας ή από 45 μέλη. Ο κύριος Λαντσπέργης λοιπόν έκανε μια προφορική τροπολογία χωρίς την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αυτή η τροπολογία του ευρωπαικου λοικου κομματος και αυτη άκυρη. Δεν σηκώθηκε το ΕΛΚ, λέει ο Πολύ συχνά συμβαίνει και δεν το καταλαβαίνω κι εγώ, λέει ο πρόεδρο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Να σας διαβάσω το άρθρο 216 του κανονισμού. Πρώτον, όταν διαπιστώνεται ένα σφάλμα σε ένα κείμενο του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος ε, συνιστά στην αρμόδια επιτροπή διόρθωση και μετά διαδίδει στο Κοινοβούλιο όταν ε, θεωρεί ότι είναι λάθος και πρέπει να λυθεί με τον τρόπο που προτείνεται. Η διόρθωση ε, κοινοποιείται τις επόμενες μέρες και θεωρείται εγκεκριμένη ε, σε περίπτωση που εντός 48 ωρών δεν διαφωνήσει η πολιτική ομάδα και δεν ζητήσει να ψηφιστεί. Σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε λοιπόν αυτού του άρθρου γιατί υπάρχει αντίρρηση στα όσα σας πρότεινα. Άρα λοιπόν θα προτείνω να ψηφίσουμε για την πρόταση αυτή. Θα διαβιβαστεί ε, στην Ολομέλεια αυτή μας η απόφαση προς ε, διόρθωση και επανόρθωση και αν διαφωνεί μια πολιτική ομάδα μπορεί να ζητήσει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Αυτό μου φαίνεται η πιο σωστή, η πιο καθαρή διαδικασία και θα σας το προτείνω να ψηφίσουμε τώρα ως εξής. Θέτω σε ψήφιση πρώτα υποστηρίζει η Επιτροπή μας να διορθωθεί η έκθεση υπέρ της διόρθωσης. Κατά. Κατά. Ομόφωνα. Ε, με μία ψήφο κατά. Χωρίς μικρόφωνο. Με μία ψήφο κατά. Ποια διόρθωση ζητάτε, λέει ο κύριος Ζατσμπέργης. Να, διαγραφεί η λέξη first. At first. Ή at first, εν πάση περίπτωση. Α, διορθώνεται την Ολομέλεια. Ε, ε, η Ολομέλεια το διορθώνει ή το Προεδρείο. Όχι, το Προεδρείο πρέπει να διορθώσουμε. Όχι, διορθώνουμε την απόφαση της Ολομέλειας. Α, αλλά ε, το Προεδρείο είναι υπεράνω όλων και αποφασίζει. Όχι, αποφασίζει η Επιτροπή μας και θα ακολουθήσουμε αυτό, διότι παραβιάστηκε ο κανονισμό. Δεν έγινε σκεμμένα, αλλά συνέβη. Τι να κάνουμε, δεν φταίει κανεί, γίνονται και τέτοια πράγματα. Ε, έγινε ένα λάθο από την Προεδρεύουσα τη Ολομέλεια. Δεν έχει ε, σημασία αν ήταν υπέρ Μάλλον δεν είχε κατατεθεί τροπολογία κατόπιν συμφωνία πολιτική ομάδα. Έχουμε διπλή παραβίαση του κανονισμού. Στην επόμενη ε, σύνοδο θα διευκρινιστεί αν δεν συμφωνεί μια πολιτική ομάδα η 40 μέλη δεν μπορεί μια προφορική τροπολογία να τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Το καταλάβαμε αυτό. Είναι σαφη θέση. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας ή όχι. Θα αποφασίσει τελικά δημοκρατικά η Επιτροπή μας ή η Ολομέλεια. Αν θα παραμείνει αυτή η έκφραση at first γιατί αυτή τη στιγμή η Επιτροπή μας προτείνει να διαγραφεί αυτό. Συμφωνώ να το διορθώσουμε το at να το κάνουμε first, να είναι και σωστά αγγλικά. Ωραία, πείστε το ΕΛΚ τότε να ε, καταθέσει και πάλι στην Ολομέλεια την τροπολογία. Αυτή είναι οι κανόνες που ισχύουν και ο κανονισμός ε, του Κοινοβουλίου και οι κανόνες γενικά είναι σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας γιατί είναι εχέγγυο και επίσης προστατεύει τις μειονότητες, τις ευάλωτες. Δεν μπορεί η συνδυπτική και μεγαλύτερη πλειοψηφία να χρησιμοποιηθεί για να παραβιάζονται οι κανόνες. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Δεν έχει σημασία η προσωπική μας άποψη. Και είναι και προπόθεση. Αλλιώ δεν μπορεί να δουλέψει ένα κοινοβούλιο χωρί κανόνε και χωρί να του στηρεί. Δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο. Και είναι σαφέστατη η θέση. Ακολουθούμε τον κανονισμό του κοινοβουλίου και όσα ορίζουν τα άρθρα τους. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει τώρα στην Ολομέλεια. Αλλά νομίζω ότι ψηφίσαμε εδώ. Μπορεί να χρειαστεί ψηφοφορία και στην Ολομέλεια. Δεν ξέρω πώς θα φτάσουμε στα αποτελέσματα. Αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις προτάσεις και έχετε πρόβλημα, υπάρχουν και άλλα ε, ένομα μέσα. Δεν τηρήθηκε ο κανονισμός. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα τι έχουμε. Μισή ώρα. Δεν ξέρω, θα έρθει νωρίτερα. But, uh, should we now make a break. Θέλετε να κάνουμε διάλειμμα ή να συζητήσουμε κάτι άλλο. Γιατί είπαμε ότι καμιά φορά θα πρέπει να συζητούμε και πολιτικά θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Και εν και της επόμενης συνεδρίασης να ακούσουμε το Συμβούλιο. Θέλετε να συζητήσουμε την παρούσα κατάσταση στο Ιράν με βάση τις νεότερες πληροφορίες για μισή ώρα μέχρι να έρθει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου. Θέλετε, συμφωνείτε. Yeah, break. Διάλειμμα. Break. A break. It's a feeling for a break. Α, θέλετε διάλειμμα, ε. Οι περισσότεροι μάλλον. Καλώς, διάλειμμα. Ο λίγων λεπτών. Αλλά να έρθει γέρος για τον Υπουργό, παρακαλώ. the ε, president of Έρχεται από το Λουξεμβούργο ο άνθρωπος που ήταν η συνεδρίαση υπουργό Εξωτερικών της Δανίας για να μας ενημερώσει και να μας αναφέρει θέματα ενδιαφέροντός μας. Να ακούσουμε τι κάνει η, η ε, δανική κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα παραδείγματα σχέσεων που έχουμε εμείς με το Συμβούλιο η Δανική Προεδρία. Λοιπόν, ραντεβού σε 20 λεπτά. Just before, if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

Κυρίε κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω στην Ομίγυρη το Δανό Υπουργό Εξωτερικό, κύριο ε, Βίλι Σεβεντάλ, σωστά το είπα. Και χαίρομαι που ήρθατε και πάλι. Είπα και προηγουμένως ότι το Συμβούλιο συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο και ήρθατε ειδικά για μας στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία που έχουμε. Και θα μας μιλήσετε εξ ονόματος κυρίας Άστο. Για ε, την, συνεδρίαση ε, του ε, Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών που συνεδριάζει για τόσες πολλές φορές. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που επανέρχομαι στην ΑΦΕΤ. Είναι το δεύτερο μου σπίτι. Χαίρομαι λοιπόν να έρθω να σας μιλήσω ε, εξ ονόματος της Κάθη Άστον ε, για τη χθεσινή συνεδρίαση. Είχαμε μία μεγάλη ημερήσια διάταξη. Μετά από τις θετικές εξελίξεις στη Βυρμανία, ακυρώσαμε τις κυρώσεις. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό να το παρατηρήσουμε γιατί ε, συνήθως επιβάλλουμε κυρώσεις. Ε, για μια φορά που χαλαρώνουμε ή αναστέλουμε τις κυρώσεις πρέπει να το πούμε. Πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση η γι' αυτό λοιπόν ε, αποφασίσαμε αυτό. Οι συμμετέχοντες ε, υπουργοί συμμετείχαν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα επόμενα βήματα στο Αφγανιστάν. Και χθε, από ό,τι ξέρω, ο κύριος άντρες ε, Ράσμουσεν, ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου, ήρθε στο Κοινοβούλιο. Του ΝΑΤΟ, συγγνώμη. Οι βασικές αποφάσεις για το Αφγανιστάν θα ληφθούν το Μάιο και το Συμβούλιο ε, σκέφτηκε τι θα γίνει με την τρέχουσα κρίση στη Συρία, ε, και στο, στην Αφρική, στο Μαλί, στην Νότια Αφρική και στην Κινέα Μπισάου. Χαιρόμαστε για τις θετικέ εξελίξεις στην Βυρμανία. Οι ελπίδες και οι προσδοκίες που εκφράζει η ΦΑΚ έχουν εκπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ε, συμφωνήσαμε λοιπόν να αναστείλουμε τις κυρώσεις εκτός από το εμπάργο όπλων και να αναθεωρήσουμε την απόφασή μας τον Οκτώβριο. Επίσης, ε, συμφωνούμε με την αξιολόγηση ότι οι αλλαγές στη Γερμανία είναι πολύ εντυπωσιακές και ειρηνικές. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ε, να εκπροσωπηθούν και οι γυναίκες της Μιανμάρ. Η κυβέρνηση κάνει πρόοδο για να υπάρξει ε, αναστολή του πυρός οι οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις επίσης προχωρούν. Οι βασικές προκλήσεις τώρα θα είναι να σταθεροποιηθεί η ειρήνη, η δημοκρατία, να υπάρξει σταθερότητα και να προχωρήσουμε ε, με τις ε, αποφάσεις για τις εθνικές περιφέρειες. Οι πολιτικοί κρατούμενοι θα πρέπει να απελευθερωθούν. Η ειρήνη που υπάρχει με τις διάφορες ομάδες είναι και οι ξένες επενδύσεις θα πρέπει να σταθεροποιηθούν. Οι υπουργοί υπενθύμησαν ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2015 και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν αλλάξει πολλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή να υποστηρίξει ενεργά την κυβέρνηση και όλους τους ενδιαφερόμενους. Η αναστολή των κυρώσεων ε, και όχι η ακύρωσή τους ε, είναι στοιχείο αυτής της πολιτικής. Είπα ότι εκπρόσωπος θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα τη Βερμανία με σκοπό να ενθαρρύνει την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και θα προσπαθήσει να βρει τρόπους για να υποστηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία με τις εθνοτικές ομάδες. Ο Επίτροπος Πίμπαξ ε, διατρανώνει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουν, ε, θα δοθούν 15 εκατομμύρια ευρώ για την ε, εκπαίδευση, υγεία και την δημιουργία δυναμικού 115 εκατομμύρια, συγγνώμη. Την τον επόμενο μήνα οι Υπουργοί Εξωτερικών θα ξανασυζητήσουν τη Βιρμανία. Το επόμενο θέμα που συζήτησαν οι Υπουργοί ήταν το Αφγανιστάν είναι βασικό... Είμαστε σε κομβική στιγμή για να προετοιμάσουμε το μέλλον του Αφγανιστάν και την ε, στάση της διεθνούς κοινότητας. Ε, η σύνδεση Κορυφής του Σικάγο το Μάιο είναι μια βασική συνάντηση, ένα βασικό ραντεβού που θα συζητήσει τη μελλοντική υποστήριξη των, εθνικών, των ε, δυνάμεων ασφαλείας του Αφγανιστάν. Στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο θα συζητηθεί η περιφερειακή κατάσταση και το Τόκιο, στο Τόκιο τον Ιούλιο επίσης. Οι υπουργοί θέλουν μια πλήρη προσέγγιση και οι τρεις αυτές διασκέψεις θα συζητήσουν ε, το μέλλον του Αφγανιστάν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ε, δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ε, ασφάλεια και τούμπαλιν. Οι υπουργοί είπαν ότι δεν αρκεί απλώς ασφάλεια, πρέπει να βρεθεί και μια πολιτική λύση στο Αφγανιστάν. Η συζήτηση έδειξε ότι υπάρχει συνένεση ε, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να παραμείνει ενεργή στο Αφγανιστάν και μετά το 2014. Είναι σημαντικό ε, ο ρόλος, υποστηρικτικό ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση για την αστυναμία και κυρίω ο ρόλο τη EUPOL για την εκπαίδευση των αστυνομικών. Το Μάιο, στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, θα δούμε ποια θα είναι η θέση τη ευρωπαϊκή Ένωση και θα υιοθετήσουμε συμπεράσματα. Μέχρι τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για υποστήριξη των ε, εθνικών δυνάμεων ασφαλείας του Αφγανιστάν μετά το 2014. Διάφοροι υπουργοί υπενθύμησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο μόνο πιθανό δωρητή και εγώ ικανοποιήθηκα που οι υπουργοί υποστήριξαν την πρωτοβουλία της ε, Δανικής Προεδρίας, το συνασπισμό των δυνάμεων, ούτως ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση των δυνάμεων ασφαλείας. Πολλοί μίλησαν έχοντας υπόψη τους τη Σύνοδο Κορυφής του Σικάγο. Μίλησαν για τη σταθερότητα του Αφγανιστάν και είπαν ότι θα πρέπει ε, γι' αυτό να υπάρξει συνεργασία με τους περιφερειακούς φορείς. Ε, ο σκοπός της συνάντησης ε, στην ε, Κωνσταντινούπολη είναι η διαδικασία της Καμπούλ. Επίσης και όλα όσα θα συζητηθούν στο Τόκιο. Οι δεσμεύσεις των δωρητών θα πρέπει να ισορροπηθούν μέσω δεσμεύσεων που θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση του Αφγανιστάν, να προχωρήσει δηλαδή με αυτά που δεσμεύτηκε στη Βόνη και νωρίτερα. Υπάρχει θέμα με την εκπαίδευση των κοριτσιών ε, υπάρχουν ανησυχίες για τον τομέα αυτό. Πάμε τώρα στην Αφρική. Ε, υπάρχουν κρίσεις σε πολλές αφρικανικές χώρες. Οι υπουργοί τόνισαν ε, την προβληματική κατάσταση στο Σαχέλ. Υπάρχει πρόβλημα με τον ανεφοδιασμό σε τρόφιμα φέτος. Οι υπουργοί συζήτησαν γενικά εκτεταμένα τη συζήτηση, στην κατάσταση στο Μαλί, που είναι αντικείμενο μεγάλης ανησυχίας. Η πολιτική κατάσταση στην πρωτεύουσα ε, δεν είναι σαφής, ενώ στα βόρεια ε, αντάρτες έχουν ε, καταλάβει τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις του Μαλί. Η ΕΚΟΜΑΣ, η οργάνωση των Δυτικών Αφρικανικών κρατών, ήταν ενεργή, ζήτησε να υπάρξει επιστροφή της ε, νόμιμης κυβέρνησης και μίλησε για μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουν την κρίση στο Βόρειο Μαλί. Ε, οι υπουργοί είπαν ότι οι γειτονικέ χώρε μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για να κρατήσουν ενωμένη τη χώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να, πει, να μείνει ενωμένη η χώρα. Εμεί θέλουμε να υποστηρίξουμε τη μετάβαση και την διενέργεια εκλογών. Αλλά θα πρέπει να το δέχεται ο πληθυσμό. Και δεν θα πρέπει να κυριαρχήσουν εκεί οι στρατιωτικοί. Οι συμφώνησαν η αποστολή της ΕΠΑ να γίνει. Θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, σχετικά έχουν υιοθετηθεί. Επίσης, οι Υπουργοί συζήτησαν της πρόσφατη βία στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν και ζήτησαν ε, να γίνει κατάπαυση του πυρός πάραφτα και οι δύο πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις και τις στρατιωτικές επιθέσεις. Ε, τα, οι διαφορές μόνο με διάλογο και πολιτική συμφωνία μπορούν να επιληθούν και όχι με πόλεμο. Η αποχώρηση χιλιάδων ε, Σουδανέζικων στρατευμάτων είναι, ήταν βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρξουν δύο βιώσιμα κράτη ε, γιατί η κλιμάκωση της βίας ε, δημιουργεί προβλήματα και αυτό ξεκαθαρίστηκε στα σύντομα συμπεράσματα του Συμβουλίου που υιοθετήσαμε σχετικά. Έπειτα, Γκινέα Μπισάου. Ε, το πραξικόπημα καταδικάστηκε και δείχνει ότι η χώρα είναι σε ευάλωτη κατάσταση και ότι οι στρατιωτικοί θέλουν να παρέμβουν. Ε, η ΕΚΟΒΑΣ αντέδρασε τάχιστα ε, και το καλωσόρισαν οι Υπουργοί, οθετήθηκαν ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου με σκοπό να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης, της ΕΚΟΒΑΣ και, τον, ε, και του ΟΗΕ. Ίσως χρειαστεί μία διεθνής εντολή βέβαια. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία συζητήθηκαν υπό τα διάφορα. Το Βέλγιο μας ενημέρωσε για την κατάσταση μετά τις εκλογές στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που γύρει λόγους ανησυχίας. Η Ισπανία έθεσε το θέμα της ε, επιδίνωσης ε, του επιχειρηματικού κλίματος στην Αργεντινή με την εθνικοποίηση ε, εταιριών ενέργειας της YPF. Η ύπατη εκπρόσωπος έκανε μία δήλωση στο Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα και η Επιτροπή Συνεργασίας θα συνέλθει που ήταν να συνέλθει μάλλον στις 20 Απριλίου, δεν ε, έλαβε χώρα. Ε, αυτές οι ισπανικές ανησυχίες ε, είναι λογικές και είπαν ότι πρέπει να, τα ευρωπαϊκά συμφέροντα να προστατευτούν. Η Ιταλία. Μίλησε για την πολιτική μετάβαση στην Ιταλία. Για τον έλεγχο των συνόρων. Για τα θέματα μετανάστευσης που θα επιδεινωθούν δεδομένοι της ε, κρίσης στο Σουδάν, Νότιο Σουδάν και Μαλή. Η Ολλανδία. Ε, μίλησε για την πρόσφατα ε, υιοθετηθής απόφαση για την, ε, για, το Σουρι... για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουρινάμ. Εγώ Μίλησα για τον Αλ Καβάχερ, ε, τον Μπαχρέιν. Φυλακίστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και εδώ και 75 μέρες κάνει απεργία πείνας. Ανησυχώ για την κατάσταση υγείας του. Ζητάμε από τον Μπαχρέιν να τον απελευθερώσει και να τον στείλει στη Δανία, γιατί είναι και δανός πολίτης. Χθες το ακαιωτικό δικαστήριο όμως α, δεν πήρε απόφαση. Θα πάρει απόφαση, υποτίθεται, μετά από μία εβδομάδα, αλλά εμείς στο μεταξύ φοβόμαστε για τη ζωή του και για την υγεία του. Όπως κάθε αρινό συμβούλιο, συζητήσαμε βεβαίως στη Συρία. Ε, και την τρέχουσα κατάσταση. Οι Υπουργοί ε, ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και Υπάρχει αυτό το ψήφισμα της UNCR και της ε, αποστολής. Επίσης, ο Κόφι Ανάν ε, θα κάνει μια αποστολή ε, με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος έξι σημείων και της κατάπαυσης του πυρός. Υπάρχουν τώρα παρατηρητές και όλοι ξέρουμε ότι είναι σημαντική η παρουσία τους το Συμβούλιο υιοθέτησε μια απόφαση για ενίσχυση των μέτρων κατά της Συρίας. Η ύπατη εκπρόσωπος μας ενημέρωσε για το Ιράν μετά την ε, πρόσφατη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τη Μέση Ανατολή και την ειρηνευτική διαδικασία εκεί, με έμφαση στην κατάσταση ε, στα κατεχόμενα στην Παλαιστίνη και συμφώνησαν να το ξανασυζητήσουν αυτό το θέμα στην επόμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών το Μάιο. Στα... Εγώ εκπροσώπησα την ύπατη ε, εκπρόσωπο στο ετήσιο Συμβούλιο Συνεργασίας με το Μαρόκο που γίνεται στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του ΦΑΚ. Αυτή είναι η παρουσίασή μου κυρίες και κύριοι. Ε, Αυτά έχω να σας πω εκ μέρους της ΥΠΑ εκπροσώπου. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ερωτήσεις, ο κύριος Αλαφράγκα. Ε, ε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό Εξωτερικών. Χαιρετίζω αυτό που είπατε, ότι αισθάνεστε εσά το σπίτι σημαίνει ότι σα φερόμαστε πάρα πολύ καλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κα... Πράγμα το οποίο δεν συμμερίζονται όλοι όσοι έρχονται εδώ να συζητήσουν μαζί μας. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Όντως, εχθές είχαμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που μας μίλησε ότι για την θέλησή του να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με ένα σχέδιο έξι σημείων. Θα ήθελα λοιπόν να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς συζητήσατε στο Συμβούλιο ε, πιο λεπτομεριακά για το Αφγανιστάν. Είπα ανήγγυλαν μια σειρά μέτρων κατά του Ιράν και της Συρίας, κυρίως ε, για το θέμα της καταστολής του κύβερνο εγκλήματος. Εσείς συμφωνείτε αυτή την ε, πολιτική επίσης ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή. Τι σκέφτεστε για την ε, ακύρωση του Συμβουλίου για το φυσικό αέριο μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ μετά την καταστροφή των διαφόρων αγωγών φυσικού αερίου, όπως ξέρετε, εξαρτάται πάρα πολύ από αυτό το Ισραήλ. Και τελικά, κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στη Ρεψόλ μετά από την εθνικοποίησή της από την κυβέρνηση Αργεντινής. Και για την εθνικοποίηση και το γεγονός που δημιουργείται από την, ε, για τους μετόχους. Το συζητήσαμε αυτό και στην Ολομέλεια. Έγιναν κάποιες σαφέστατες δηλώσεις και εκ μέρους της ε, ε, ε, εκπροσώπου. Δεν είδα όμως κανένα διατάφτα εκ μέρους του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε το Συμβούλιο πώς αντιμετωπίζει αυτή τη μεγάλη ανησυχία που εκφράστηκε εκ μέρους της κυβέρνησής μας και ποιες είναι οι θέσεις και αν η τοποθέτηση του Συμβουλίου σχέση με το θέμα αυτό. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω προς το παρόν κύριε Πρόεδρε και πάλι σας ευχαριστήσω την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Thank uh, Κύριε Γκόμες. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε και εγώ να ερωτήσω το εξή τον Προεδρεύοντα. Πιστεύετε ότι θα έχουμε εκ μέρου των αρχών της Βερμανίας κάποιες διασφαλίσεις ότι θα μπορέσουν να στείλουμε το προσωπικό που χρειάζεται για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το πρόγραμμα το οποίο έχει προβληθεί. Η Lady Ashton θα φέρει επιστρέφοντας και αυτές τις διασφαλίσεις και θα υπάρξουν και εγγυήσει ότι οι πολιτικοί ε, κρατούμενοι θα ελευθερωθούν και θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι θεμελιώδεις διδικήσεις όπως τις ελευθεροτυπίες μεταξύ άλλων. Όσον αφορά το Αφγανιστάν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. σε σχέση με τους ε, φορείς οι οποίοι αντίσουν δραστηριότητε σε εκείνη την περιοχή. Ποια είναι οι επιπτώσεις της χρησιμοποίησης των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Είναι κάτι το οποίο με αυτά τα οποία συνέβησαν δημιούργησε ένα πάρα πολύ αρνητικό προηγούμενο γενικότερα, αλλά νομίζω ότι οι επιπτώσεις ήταν δραματικές κυρίως στις γειτονικές χώρες για το Πακιστάν. Άκουσα ότι καλής μπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο αεροσκάφος για 300 δολάρια. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα δεδομένου ότι είναι σοβαρό το θέμα. Όσον αφορά την Αφρική, χαίρομαι για αυτά τα οποία είπατε. Κυρίως μιλήσετε για την ε, Λιβύη και πρέπει να δούμε, όπως είπατε και εσείς, τι σημαίνει στο Μαλί, στην Κινέα Μπισάου και τις επιπτώσεις ε, για το ε, Σουδάν με τη Λιβύη. Θα στέλνω να σας ερωτήσω. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει τη Λέιδη Άστον, ώστε να υποστηρίξουμε με τον κατάλληλο τρόπο την ανάπτυξη ε, και την αποστολή αντιπροσωπεία στη Λιβύη. Ξέρω ότι ε, μια ήδη υπάρχουσα αντιπροσωπεία επιστρέφεται, αλλά θα πρέπει να ε, στείλουμε κι άλλη αντιπροσωπεία, κυρίως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο Μπενγκαζί, δεδομένου ότι υπάρχουν επιπτώσεις και για τη Λιβύη και για μας Τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει η θέση σας για την Guinea-Bissau, για την καταδίκη των συμβαίνουν, για την απελευθέρωση των φυλακισμένων. Άκουσα όλα αυτά, αλλά δεν βλέπω κάτι το οποίο θα είναι πρωταρχή σημασία την άποψή μου. Δηλαδή, να υπάρχει μια αντιπροσωπεία ε, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας στην Κινέα Μπισάου. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, απαραίτητο για να έχουμε τις αποδείξεις ότι πρόκειται για μια πραγματική ε, κυβέρνηση και ένα κράτος που λειτουργεί σωστά και όχι κάποιον ο οποίος κρύβεται πίσω από όλο αυτό το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Είναι σημαντικό λοιπόν όλα αυτά να μπορέσουμε να τα κύριε Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Για την Αργεντινή. Νομίζω ότι αναφέρατε το πρόβλημα αυτό της ε, εθνικοποίησης της ε, Ρεψόλ από την πρόεδρο Κίρσον και υπάρχουν πολλές πιέσεις προς τις ξένες τράπεζες, κυρίως τις αγγλικές οι οποίες τις δραστηριότητε στην Αργεντινή. Εάν θέλουν να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα πετρελαίου κυρίως στα νησιά Φόκλαν. Ξέρετε πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός από την Ισπανία, ποιες άλλες χώρες είναι αυτές, ποιες είναι οι χώρες που υποστηρίζουν αυτό το οποίο ε, υπάρχει ως πρόβλημα μεταξύ της ε, Αργεντινής και των νησιών Φόκλαν. Το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο θίξατε στις συζητήσεις σε σχέση με την ε, ε, εθνικοποίηση που έγινε εκ μέρους της Αργεντινής και των αντισταθμισμάτων ενδεχομένως θα δοθούν στην κυβέρνηση της Ισπανίας. Όπως ε, ε, βλέπουμε, αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται αυτή η κυβέρνηση όσον αφορά και τα θεμελιώδη και βασικά δικαιώματα και με την απαλωτρίωση ιδιωτικής ε, ιδιοκτησίας. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα των πολιτικών κρατουμένων και της, ε, των ε, κυβέρνησης στο Μπελαρούσου. Επίσης, το θέμα στην Ουκρανία που έχει δημιουργηθεί με την ε, κράτηση της ε, πρώην Προέδρου Λουτσένκο. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα δούμε με σαφήνεια. Δεν μπορούμε σε θέματα δικαιοσύνη να είμαστε επιλεκτικοί. Δεδομένου ότι βλέπουμε κάποιοι εκπρόσωποι πρώην κυβερνήσεων να βρίσκονται σε διαρκή δίωξη. Τώρα, όσον αφορά την Ρωσία τη νέα κυβέρνηση Πούτιν. Πιστεύετε ότι ο τωρινός πρόεδρος Πούτιν θα είναι πρόεδρος μάλλον των μεταρρυθμίσεων και θα προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο να κάνει ένα κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα που φοβούμε ότι βρίσκεται σε διαρκή ε, πόλεμο και εξισορρόπηση μεταξύ κράτους και κλεπτοκρατών. Επίσης, το θέμα αυτό που δημιουργείται με τον, τον θάνατο του κυρίου Μαγνίσκη, ε, ε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, τι ακριβώς έχετε να μας πείτε για την Ευχαριστώ. Κύριος Μέγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που κάνετε. Καταλαβαίνω ότι στη συζήτηση του Συμβουλίου Ίσως δεν συζητήσετε επιτομερικά το θέμα της πολυεθνικής όπως η Ρεψόλ. Δεν διαφωνώ, διότι πιστεύω ότι τα προβλήματα που έχει μία πολυεθνική δεν έχουν μεγάλη σχέση με την ημερήσια διάταξη την οποία εσείς συζητήσατε. Αρχίζω από το Σάχελ, πρέπει να σας πω ότι εμένα με απασχολούν περισσότερο τα 10 εκατομμύρια άτομα τα οποία εξαιτία του προβλήματος του οποίου υπάρχει αύριο θα πεθάνουν διότι δεν έχουν να φάνε. Και το θέμα το ελάχιστου ποσοστού της επιστηστικής βοήθειας των όλων αυτών των εκατομμυρίων που φτάνουν στα χέρια τους. Είναι λοιπόν επαρκές αυτός που γίνεται και αν δεν κάνουμε κάτι ε, ε, γρήγορα θα πεθάνουν οι περισσότεροι. Από τις 8 χώρες του Σαχέλ στις 7 υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Τώρα, το θέμα της πολυεθνικής είναι θέμα πείνας και κανένας μέτοχος δεν θα πεθάνει. Κανένας. Κατά συνέπεια, χαίρομαι που δεν το συζητήσετε αυτό το θέμα. Και αν τέτοιου είδους θέματα που θέτουν σε αμφισβήτηση τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι εννοούν τις ε, σχέσεις ανά τον κόσμο, δεν θα πω ότι συμφωνώ. Χθε ο κύριος Ρασμούσεν, εκ μέρου των άτομων, μα είπε ότι δεν θα πρέπει να αποφεληθούμε από την κρίση για να ε, μειώσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Περού αυτού όμως πρόκειται. Το σημαντικό είναι να μειώσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Πώς είναι δυνατόν όλα τα κονδύλια που πηγαίνουν για την κοινωνική πολιτική στην Ευρώπη να μειωθούν και να μην μειώνονται τα κονδύλια που πάνε στις αμυντικές δαπάνες. Πώς είναι δυνατόν να μην βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ όλων και να μην θέτουμε σε πρακτική εφαρμογή ε, αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν στην ε, ατζέντα της ε, χιλιατίας. Αυτό εμάς μας απασχολεί. Και θα θέλαμε η, το ΟΗΕ να δώσει τα κατάλληλα κονδύλια για να μπορέσει το δράμα αυτό της ανέχειας και της πείνας να μπορέσει να επιληθεί. Τώρα, Φαίνεται ότι σε σχέση με το Ιράν. Από ό,τι ακούσα από το ταξίδι της κυρίας Στάστον, δεν υπάρχει πρόβλημα για να μπορέσουν ε, να επισκεφθούν οι διάφορες αντιπροσωπείες που θέλουμε, τις ε, εγκαταστάσεις πυρηνικές. Βεβαίως κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι χρησιμοποιεί για ειρηνικούς λόγους ε, το Ιράν την πυρηνική ενέργεια μόνο. Θα πρέπει όμως να μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε και θα πρέπει να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για να επαληθευτούν κάποια πράγματα και να μην ακούσουμε μόνο τι έχει να πει το Ισραήλ με τις κατηγορίες του και ξαναγυρίσουμε πίσω σε τέτοιου είδους παλιές ε, σχέσεις που είχαν στο παρελθόν ε, στην περιοχή. Βεβαίως έχει και στη διάθεση του πυρηνική ενέργεια τη χρησιμοποιεί το Ιράν. Κανένας όμως δεν κούνησε ούτε το παραμικρό ε, από την κατάσταση εκείνη για να διδαχθεί. Τώρα, σε σχέση με την ε, πρόβλημα το οποίο υπήρχε στη, με το Μαρόκο και την ε, δυτική περιοχή της Σαχάρας. Πρέπει να πω ότι ακούστηκε ότι το Μαρόκο τώρα τελευταία στην περιοχή αυτή κατασκοπεύει εκ μέρους του ΟΗΕ. Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία ώστε να εγγυηθούμε ότι όχι μόνον ε, μπορούμε να ε, εποπτεύσουμε την όλη κατάσταση όσον αφορά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά να χειριστούμε και το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Λόχ Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ήταν μακρά ε, η ημερήσια διάταξη, αλλά παρόλα αυτά ε, χαίρομαι που πήρατε πρωτοβουλία για να υπερασπιστείτε το πολιτικό κρατούμενο στον Παχρέν που κάνει και απεργία πείνας. Για τη Βυρμανία στο Κοινοβούλιο εγκρίναμε ένα συνολικό ψήφισμα ε, που σκιαγραφεί και όλα τα προβλήματα εκεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά όπως σας είπα, τώρα εσείς έχετε αναστείλει τις κυρώσεις. Και έχω καταλάβει ότι ορισμένοι στρατιωτικοί που δεν είναι ακριβώς μεταρρυθμιστές στη Βυρμανία ελέγχουν ακόμα την ξυλία ε, και τη βιομηχανία. Ε, τις κυρώσεις, αν τις άρετε όχι σταδιακά αλλά συλλήφθην και κατευθείαν, πώς θα επιβεβαιωθείτε ότι δεν θα υποφελούνται οι λάθος άνθρωποι. Αυτή ήταν ερώτηση και μία σύσταση. Ακούμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για δυνατότητες, για ε, ε, τις εξωτερικές σχέσεις, για το Υπουργείο Οικονομίας. Χρειάζεται να δημιουργηθούν θεσμοί εκεί, σχεδόν σε όλους τους κλάδους της πολιτικής. Ακριβώς λόγω της απομόνωσης πιστεύω ότι οι φοιτητέ από τη Βυρμανία δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα Erasmus Mundus. Και θα ήθελα να παρακαλέσω την ύπατη εκπρόσωπο να το κοιτάξει αυτό και να βρει έναν τρόπο, μια ειδική ρύθμιση για να έχουν εκπαίδευση και κατάρτιση φοιτητέ από τη Βυρμανία και πράγμα το οποίο θα τους ικανοποιήσει πάρα πολύ και θα εκτιμήσουν. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Και μετά θα κάνουμε και άλλο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ για τον κύριο Σαλαφράνκα για το Αφγανιστάν. Είναι τέσσερα τα ζητήματα που θα καθορίσουν το μέλλον του ε, Αφγανιστάν. Το πρώτο είναι η ασφάλεια. Διότι χωρίς ασφάλεια, ό,τι και να γίνει θα καταργηθεί, θα ακυρωθεί. Ούτε παιδεία μπορείς να εξασφαλίσεις, ούτε γυναικεία δικαιώματα, ούτε ανάπτυξη, οποιασδήποτε δυνατότητα στη χώρα, χωρίς ασφάλεια. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό. Δεύτερο σημαντικό είναι η προθυμία να συνεισφέρουμε σε αναπτυξιακή βοήθεια για πολλά χρόνια προς τη χώρα, γιατί δεν θα είναι οι ίδιοι σε θέση να το κάνουν μόνοι τους για τα επόμενα χρόνια. Το τρίτο να βοηθήσουμε να ενισχυθεί η αφγανική οικονομία. Και επιστημιστικός κλάδος, τα τρόφιμα, οι δυνατότητες μεταφορών. Η εξορρυκτική βιομηχανία ενδεχομένω και άλλα. Για να μπορέσει το Αφγανιστάν να ορθοποδήσει. Και το τέταρτο σημαντικό είναι τα γειτονικά κράτη. Χώρες όπως το Πακιστάν βεβαίως και το Ιράν, η Ρωσία, η Ινδία. Ποιο ρόλο θα διαδραματίσουν οι χώρες αυτές εκεί. Και νομίζω ότι και τα τέσσερα αυτά θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Και ένα πέμπτο, χωρίς αυτό είναι λιγότερο σημαντικό, είναι το πώς θα διαμορφωθεί η εσωτερική πολιτική σκηνή στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει να γίνουν πολλές συμφωνίες, θα πρέπει να γίνουν ε, πολλές ε, συμβαστικές ρυθμίσεις και να συμπεριληφθεί πολλοί κόσμος στο πολιτικό γίγνεσθε. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα γυναικεία δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών και η εκπαίδευση ε, των παιδιών και τα σχόλια είναι πολύ σημαντικό. Ρωτήσατε και για τη Μέση Ανατολή για τον αγωγό φυσικού αερίου και τις επιθέσεις που δέχτηκε. Βεβαίως είναι πολύ ανισχυτικό. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου η ασφάλεια έχει χαλαρώσει, έχει αποδυναμωθεί στην περιοχή. Και αυτό δείχνει την ανάγκη εξέβρεσης λύσης μέσα από διαπραγμάτευση για την περιοχή γενικότερα. και αν μπορούσα να δώσω μια καλή συμβολή στους Ισραηλινούς, είναι ότι έχει έρθει η ώρα να σκεφτούν σοβαρά την πολιτική συμφωνία και προς όφελος του ιδίου του Ισραήλ, αλλά και προς όφελος των Παλαιστινίων. Μπορεί να είναι η τελευταία γενιά που είναι διατεθειμένη να κάνει πολιτική συμφωνία. Γιατί τώρα βλέπουμε, μετά από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων, ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί πολιτική λύση αυτή καθ' αυτή. Και όποιο αγαπάει και τις δύο χώρες παρακαλώ να τους πει να πάρουν σοβαρά υπόψη τους. Αυτό τελειώνει ο χρόνος για τη δυνατότητα που υπάρχει εξέβρεση πολιτικής λύσης και μετά από διαπραγμάτευση. Τώρα, για την εθνικοποίηση τη εταιρεία ε, ε, EPF. Ότι αν θέλει κανεί να εθνικοποιήσει μια εταιρεία μπορεί να το κάνει αλλά ακολουθεί κάποιους κανόνες. Υποστηρίχθηκε αυτό από τους Ισπανούς, αλλά ε, θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Θα πρέπει να μας εξηγήσει η Ισπανία τι προτίθεται να κάνει για τη Συρία. Νομίζω Αν υπάρχει κάτι θετικό, σήμερα είναι οι παρατηρητές, οι οποίοι θα κάνουν διάφορα πράγματα. Θα αναφέρουν στον κύριο Ανάν και στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το τι συμβαίνει στη Συρία. Επίσης, ενδέχεται να δούμε ε, το, την ίδια κατάσταση που ε, διαπιστώσαμε όταν ήταν και ο Αραβικό Σύνδεσμο, ότι τολμάει ο κόσμο ξαναβγαίνει στον δρόμο και να διαδηλώνει, γιατί αισθάνονται κάπως ότι τους προστατεύουν. Όπως και οι δημοσιογράφοι μπορεί να θεωρήσουν ότι προστατεύονται από την παρουσία των παρατηρητών και να βγουν και να γράψουν και εκείνοι τι συμβαίνει. Επίσης, άλλο σημαντικό είναι ότι συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας από όλα τα μέλη του που σημαίνει ότι στο εξή και η Ρωσία και η Κίνα δεσμεύονται και δεν μπορούν να παραμείνουν παρατηρητές ή αν επιστρέψουν οι παρατηρητές και πούν ότι δεν έχει γίνει τίποτα από τα βήματα που προτείνει το σχέδιο ανάν. Σύντομα για την Αφρική και απαντώ σε πολλούς από εσά που με ρωτήσατε. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικά τα όσα συμβαίνουν. Είναι πραγματικά πολύ άσχημη η κατάσταση. Πήγα εκεί εξ ονόματος ε, της κυρίας Άστον στο κέρας της Αφρικής ε, πριν από δύο εβδομάδες και στην Ιγυρία πριν από δύο μήνες. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι αυτό το μείγμα φτώχειας, βαθιά ανησυχητικής ένδυας, όπως είπατε και εσείς κύριε Μάγερ, αλλά ταυτόχρονα και αυτά τα δύο συνδέονται, αναδύονται νέες τρομοκρατικές ομάδες που ενδέχεται να συνδέονται ε, μεταξύ τους Πόκο Χάρεμ ε, στη Βόρεια Νιγηρία και η Αλκάιντα επίσης ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική καταστροφή που κινδυνεύει να επέλθει ε, αν δεν αντιδράσει κανείς. Είναι σημαντικό να είμαστε παρόντες, να βοηθούμε την ΕΚΟΒΑΣ που είναι η οργάνωση των κρατών της Δυτικής Αφρικής που πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και προσπαθεί να βοηθήσει στην περιοχή. Το θετικό ποιο είναι στην Αφρική πέρα από όλες τις ε, άσχημες ειδήσει είναι ότι οι Αφρικανοί ηγέτες, οι Αφρικανικές χώρες αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι ίδιοι για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις. Όταν πήγαμε στην Αντίσα Μπέμπα, στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, ε, Μάλλον, ε, όταν ήμασταν στην Αντισαμπέμπα ε, γινόντουσαν διαπραγματεύσεις του, του Σουδάν με τον Νότιο Σουδάν στο ίδιο ξενοδοχείο που μέναμε, υπό την ηγεσία του πρώην ε, Προέδρου της Νότιας Αφρικής, του κυρίου Εμπέκη. Οπότε, ε, αναλαμβάνουν τι ευθύνες τους και θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Για τη Λευκορωσία, Ουκρανία και Ρωσία. Ανησυχούμε πάρα πολύ για τις εξελίξεις στη Λευκορωσία. Ε, έχουν αφήσει ελεύθερους δύο κρατουμένους μεν, αλλά η όλη κατάσταση είναι πολύ ενισχυτική. Από ευρωπαϊκής πλευράς έχουμε επιβάλει κυρώσεις στη Λευκορωσία, ορισμένες από τις μεγάλες τους εταιρείες και τους ε, πολιτικούς αρχηγούς. Σε ό,τι αφορά την ε, Ουκρανία, γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται με την υπόθεση της κυρίας Δημοσέγκο Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν υπογράψαμε τη συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία ακόμα και θα περιμένουμε. Τεχνικά έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις, αλλά δεν πρόκειται να υπογραφεί η συμφωνία αυτή μέχρι να επιτευχθεί πολιτική πρόοδος στην Ουκρανία. Με ρωτήσατε επίσης για το αν θεωρώ τον Πούτιν μεταρρυθμιστή. ε, δεν είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω το όνομά του. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν κάποιες ενθαρρυντικές εξελίξεις μετά τις εκλογές. Ο κόσμος τόλμησε να βγει να διαδηλώσει. Οι βουλευτικές ε, εκλογές έγιναν, ε, πρόεκυψε το αποτέλεσμα, ασκήθηκε πίεση. Παρ' όλα αυτά ε, ο κόσμος διαδηλώνει και συμμετείχε στις εκλογές. Και αυτό είναι κάπως η θετική εξέλιξη της υπόθεσης των εκλογών. Αλλά τώρα νομίζω ότι ο Πούτιν θα ε, κυβερνήσει τη Ρωσία με τον τρόπο που ξέρουμε και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ομάδες αντιπολίτευσης. Έχουμε επαφές μαζί τους και βεβαίως έχουμε επαφές και με τους Ρώσους πολιτικούς γενικότερα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και ίσως σε 20-30 χρόνια να έχουν μια πιο ζωντανή δημοκρατία. Ε, το ελπίζω. Α, για τη Βερμανία, για να τελειώσουμε αυτό. Ε, τρεις είναι οι βασικοί ισχυρισμοί τους. Ο πρώτος είναι ότι οι εκλογές της 1ης Απριλίου δεν εξήχθησαν πάρα πολύ καλά όπως θα ελπίζαμε και ελπίζαμε. Το δεύτερο είναι η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Έχουν αφήσει ορισμένους ελεύθερους, αλλά περιμένουν κι άλλοι. Και το τρίτο που θέλαμε είναι οι μειονότητες να προστατεύονται. Υπάρχουν ακόμα εντάσεις και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό. Αυτά τα τρία λοιπόν θέλαμε από τη Βυρμανία. Εγώ προσωπικά είμαι λίγο αισιόδοξο. Έχουν λάβει μια στρατηγική απόφαση ε, και οι στρατιωτικοί το έχουν καταλάβει, θέλουν να είναι ένα μέρος του κόσμου. Μπορεί να σφάλω. Εμείς μπορεί να ε, αναστήλαμε τις κυρώσεις. Αναστολή σημαίνει ότι μπορούμε να τις επαναεπιβάλλουμε αν υπάρξει στρεβλή εξέλιξη. Πάντως, Τώρα συνεχίζεται ε, αυτή η ε, αντιπαράθεση μεταξύ των προνομιούχων που είχαν την εξουσία και εκείνων που δεν είχαν την εξουσία, το μη προνομιούχων. Έχουμε πολιτικές επαφές με ομάδες και της Βυρμανίας και προσπαθούμε και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουμε την πολιτική διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλα τέσσερα άτομα θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Σας ζητώ να περιοριστείτε ο καθένας ένα λεπτό Κύριε Πρέντα, παρακαλώ, ακούμε την ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Θα κάνω ένα σχόλιο για τη σημασία που δίνετε στην Αφρική. Σας ευχαριστώ που ήρθατε βέβαια μαζί εδώ και μας μιλήσατε σήμερα. Θέλω να σταθώ λίγο στην κατάσταση στο Μαλί, γιατί είναι μια λεπτή κατάσταση εκεί. Το Μαλί μέχρι πρόσφατα ήταν ο καλός μαθητής της τάξης. Ο πρώην πρόεδρος ήταν ένας από τους ε, λίγους πρόεδρους της Αφρικανικής Υπήρου που είχε έρθει όχι μόνο στην Επιτροπή μας αλλά και στην Ολομέλεια να μιλήσει και βάλατε το θέμα της στόχιας ε, και της ε, ανάδυσης νέων θυλάκων τρομοκρατίας πολύ σωστά. Επίσης, ο στρατός είναι πολύ ασθενής, είναι πολύ δραματική η κατάστασή του και αυτό μπλοκάρει την επίλυση του προβλήματος του Βορρά και δεύτερον η διένεξη με τους γείτονες, κυρίως με τη Μαυριτανία. Έχουν διαφορετική στρατηγική στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ε, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση τώρα που ο πρόεδρος της Μαυριτανίας ε, αποδυναμώθηκε από τις διαμαρτυρίες του Ισλαμικού κόμματος που έγιναν πρόσφατα. κυρία Λόπες, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση. Η ερώτησή μου έχει σχέση με το Μαλί. Σε σχέση με τον ρόλο που διαδραματίζει η γερία στην περιοχή. Όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα της κοινότητας του Αρέγγι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην διάνεξη αυτή και η ρόλος που μπορεί να παίξει η Αλγερία είναι ρόλος αποσταθεροποίησης είστε ενήμερο για τέτοιου θέματα, διότι όντω οι ομάδες Αλκάδια, ε, της Αλκάιντα έχουν την... Έλκουν, προέρχονται από την Αλγερία. Έχετε πληροφορίε για τι τις μυστικές υπηρεσίες της Αλγερίας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για το ρόλο της στην αυτή. Ευχαριστώ, κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, σας άκουσα με ενδιαφέρον από την ανακοίνωση τύπου για το Συμβούλιο Βλέπω ότι μιλήσατε για την ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή και τις πυρηνικές συνομιλίες για το Ιράν, για το Ισραήλ, πρωτόκολλο συμφωνία σύνδεξης και πάλι για το Ιράν, περιοριστικά μέτρα. Εκπλήσουμε πάρα πολύ. Το θέμα αυτό είναι πρωτοσέλιδο κάθε μέρα στον Ισραηλινό τύπο και εκεί δεν έχετε αποφανθεί για την ενδεχόμενη επικείμενη επίθεση του Ισραήλ και το βομβαρδισμό ε, πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Σας ρώτησε και ένας συνάδελφος, εσείς δεν απαντήσατε νομίζω. Έχουν άποψη οι υπουργοί γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει στεναρή θέση σχετικά. Αν κάθε μέρα πάει και ένας άλλος υπουργός εκεί και το σητάει και είναι έτοιμοι να επιτεθούν να το συζητάμε κι εμείς ε, και να λέμε καθημερινά ότι δεν το θεωρούμε καλή ιδέα. Τι λέει το Συμβούλιο γι' αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει κυρία Ντεκαϊζέρ. Τρεις ερωτήσεις. Για τη Συρία Λίβανο είναι η πρώτη. η κατάσταση της Συρίας στο, και η επίπτωσή της στο Λίβανο είναι πάρα πολύ σημαντική και πολιτικά και ανθρωπιστικά. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στους πρόσφυγες. Ε, υπάρχει κανένα θέμα, καμιά συζήτηση για το Λίβανο, για το Σουδάν, Νότιο Σουδάν. Κατά τη διάρκεια της ε, ανεξαρτησίας του Νότιου Σουδάν, εμείς και οικονομικά συνεισφέραμε και επιμελητιακά. Ε, αλλά μετά το ξεχάσαμε το Σουδάν. Ενώ ξέραμε ότι το πρόβλημα δεν είχε επιληθεί. Είχαμε πολλές ελπίδες και δώσαμε και πάρα πολλά λεφτά ε, στην ομάδα υψηλού επίπεδου του Ελμπεκή για να επιληθούν τα εκκρεμή προβλήματα, ιδίω ε, πώ θα μοιραστεί το πετρέλαιο κτλ. Τελικά υπάρχει μια αξιολόγηση του τι συνέβη, γιατί ξαφνικά εμφανίζεται στο, στην ατζέντα μας το Σουδάν. Ε, κάναμε τις καλές επιλογές, τις σωστές επιλογές. Και τρίτο και σύντομο. Στο τέλος των συμπερασμάτων σας αναφέρατε ότι στη σχέση μας με το Ισραήλ έγινε μια ανταλλαγή επιστολών για να τροποποιηθεί το, τα παραρτήματα του πρωτοκόλλου 1 και 2. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα από αυτά που λένε τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Προεδρεύοντα, μάλλον. Ευχαριστώ. Για το Μαλί πρώτα απ' όλα. Υπάρχει κίνδυνος η κατάσταση αυτή να έχει επιπτώσεις και στις γειτονικές χώρες. Θα πρέπει λοιπόν, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε εκ νέου θέσεις, ε, ε, σχέσεις σωστές μεταξύ του Μαλή και των γειτονικών χωρών. Και βεβαίως να ληφθεί υπόψη η κατάσταση στην Νιγηρία. Ηνωμένα Έθνη θα λάβουν τα απαραίτητα μέσα νωρίτερα από ό,τι αναμένεται στην περιοχή του Σαχέλ για να μην υπάρξουν καταστάσεις πιο επικίνδυνες. Ξέχασα να απαντήσω μια ερώτηση από πριν. Στην Λιβύη, τέτοια κατάσταση, αυτοί οι οποίοι ήταν υπέρ του Καντάφη μετακινήθηκαν νοτίως με τον οπλισμό που διέθεταν και δημιουργούν κάποιες εντάσεις και βεβαίως οι ένοπλες διενέξεις είναι πιο επικίνδυνες από άλλες. Όσον αφορά την αναμενόμενη επίθεση του Ισραήλ προς το Ιράν. Πάρα πολλές φήμες υπάρχουν περί του θέματος. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων στα οποία θα οδηγηθεί η Λέιδη Άστον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι όπως το τι γίνεται σε επίπεδο πρωταθλήματος για ωραίες φορές για στο ποδόσφαιρο πολλά. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς βεβαίως δεν είμαστε κύριοι παίκτε σε σχέση... Which could be of great importance uh, for us. Ή οι μεγάλοι σατανάδες ή οι μεγάλοι κακοί όπω είπα σε αυτή την περίπτωση. Πιστεύω λοιπόν και αυτή την προσωπική μου ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εάν υπάρξει επίθεση. Διότι υπάρχει κίνδυνος γενικότερης έκρηξης στη Μέση Ανατολή, η οποία θα είναι ανεξέλεγκτη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι ό,τι κάνουν τώρα ε, για να ευρεθεί μια λύση μετά από διαπραγμάτευση και σε επίπεδο δικό μας και σε επίπεδο ΙΟΙΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως το Ιράν, όπως και πολλές άλλες χώρες που διαθέτουν πυρηνική ενέργεια, μπορούν να έχουν το δικό τους πρόγραμμα για τη χρήση της, για, τη χρήση σε ειρηνικούς, για ειρηνικούς σκοπούς. Βεβαίως δεν ε, έχει το δικαίωμα να αναπτύξει πυρηνικό πλεισμό και χρησιμοποιήσει γι' αυτό το λόγο την πυρηνική ενέργεια. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το θέμα των προσφύγων στον Λίβανο. Όπως ξέρετε, μέρος της Συρίας. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες και πολλοί πηγαίνουν και προς την Τουρκία. Προβλέπουμε για τους πρόσφυγες αυτές και στις χώρες αυτές ε, οικονομική βοήθεια για να βοηθήσουμε τις χώρες που δεν διαθέτουν τα κονδύλια και κάνει και η Τουρκία κάποια στρατόπεδα υποδοχής προσφύγων, δίδονται πολλά ποσά και νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες αυτές οι οποίες υφίστανται τον μεγάλο φόρτο αυτό προσφύγων. Τώρα σαν αφορά το Σουδάν. Οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα υπό την ηγεσία του πρώην Πρόεδρου της ε, Νοτιοαφρικής και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να επιτύχουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και, το, πώς είπαμε, το κράτος του ε, Νοτίου Σουδάν έχει δημιουργηθεί. Το θέμα των ορίων των δύο χωρών είναι ακόμη κρεμές και βεβαίως υπάρχει το θέμα της μεταφοράς του πετρελαίου προς το κύριο λιμάνι. Και υπάρχει και το θέμα των μειονοτήτων. Το θέμα λοιπόν αυτό θα πρέπει να επιληθεί υπό την αιγίδα της οργάνωσης που είναι η καλύτερη και πλέον καταρτισμένη για να μπορέσει να λύσει αυτό το πράγμα. Και αυτό γίνεται και με την συνδρομή της, του πρώην Προέδρου της Νοτιοαφρικής. Yeah. Okay. I forgot uh, να απαντήσω και σε μία ερώτηση για τα θέματα της ΕΠΑ στην Κινέα Μπισάου. Τώρα θα σας απαντήσω λοιπόν. Πριν από ένα χρόνο σταμάτησε νομίζω γιατί δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης των στρατιωτικών και έτσι οποιαδήποτε συζήτηση για αυτά τα θέματα σταμάτησε. Δεν θα αποφασίσουμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση σε θέματα πολιτικής. Ε, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα αποκατασταθεί η κατάσταση στην Κινέα Μπισάου και θα έχουμε βεβαίως ε, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την τόσο ε, ευάλωτο και, ε, ευάλωτο και ασθενές κράτος αυτός. Πιστεύω ότι μάθαμε από αυτά τα οποία συνέβησαν πρόσφατα. Δηλαδή, πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε καλύτερο σχεδιασμό ώστε να υπάρξει πιο λειτουργικό και καλύτερο κράτος διακυβέρνησης στην ε, Γκινέα Μπισάου. Αυτά είχα να πω προς παρόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θέλει κανείς να προσπαθήσει κάτι. Πολύ σύντομο κύριε Στέμις. Θα έπρεπε να την αγροτήσει αυτό, αλλά ξέχασα. Στον τύπο καλύφθηκε πάρα πολύ ε, από εμάς το τι ακριβώς γίνεται στην Κίνα, στη μεγάλη ε, μάχη αυτή που διεξάγεται σε επίπεδο κόμματος με αυτή την ε, δολοφονία του Άγγλου υπηκόου και ενδεχομένως τη δολοφονία και ενός Γάλλου υπηκόου από την κυρία αυτή συζητήσατε ε, εσείς αυτό το θέμα, το τι ακριβώ γίνεται σε επίπεδο ηγεσία Κομμουνιστικού Κόμματο της Κίνας. Γίνεται τίποτα σε επίπεδο σχέσεων. Τι ε, γίνεται με αυτούς οι οποίοι δολοφονούν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συζητήθηκε αυτό το θέμα χθε, αλλά ξέρουμε ότι θα υπάρξουν η νέα ηγεσία στην Κίνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια κινέζικη ηγεσία η οποία με θάρρος θα προχωρήσει σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς. Βεβαίως, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, δεν ξέρουμε τίποτε, δεν είμαι σε θέση λοιπόν να σας απαντήσω σε αυτές τις συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, που μου κάνετε. Δεν έχω ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο και μπήκατε στον κόπο να έρθετε να μας ενημερώσετε και σας εύχομαι καλή συνέχεια ε, και καλή συνέχεια στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ και καλή επάνωδο στη θαυμάσια Κοπενχάγη. Και ξέχασα να αναφέρω και τον Πιέρεμον που ήρθε και πάλι και ήταν παρόν και εκείνος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω το επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης. Είναι κοινή συζήτηση, παρουσία εμπειρογνωμών. Όχι με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή. Με θέμα την οδηγία για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, οδηγία της Επιτροπής. Αν μπορεί κάποιο να βάλει λίγη διαφάνεια στον τίτλο τον ίδιο και μετά στην υπόλοιπη έκθεση. Θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Και με μεγάλη χαρά Σας ανακοινώνω ότι έχουμε τις δύο γνωμοδοτήσεις προς την Επιτροπή ε, Ελευθεριών και την Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων. Έχουμε και κάποιους εμπειρογνώμονες, όπως είπαμε, ενώπιον μας. Για να τους ακούσουμε. Χρόνο δεν έχουμε πολύ όμως. Τέσσερα λεπτά έκαστος εμπειρογνώμων και μετά η κυρία Μπραντνερ θα μας εξηγήσει τι είπαν οι εμπειρογνώμονες. First, I would like to give the floor to... Καταρχάς, να δώσω το λόγο στην κυρία Σελιχάν. Ορίστε. Που ήταν ε, επικεφαλής των συμβούλων του, στο γερουσιαστή Κάρντιν για την αντίστοιχη πρόταση ε, που τελικά Dot Dodd-Frank Act. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να μιλήσω το, για το 1504 και να συζητήσω για τις επιπτώσεις ε, στις οδηγίες αυτής, αυτές περί διαφάνειας. Είναι ιστορική αλλαγή για, την, για τον κλάδο και για την κυβέρνηση και ελπίζω να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στο, στις χώρες. Θα ήθελα να εστιάσω σε δύο βασικά θέματα που είναι σημαντικά για τη συζήτηση και για το πώς εφαρμόζουν οι αρμόδιες επιτροπές το νόμο στις ΗΠΑ και για το πώς αυτό εσάς ενδιαφέρει. Ε, έχουμε τον νόμο τα, οι συνολικές ε, για κάθε τέτοιο project της εξορρυκτικής βιομηχανίας. Έχουμε την υποχρέωση να λογοδοτήσουμε, να συντάξουμε εκθέσεις. Επίσης, ε, η Επιτροπή α, της Κεφαλαιαγοράς ε, έχει έρθει, έχουμε έρθει σε επαφή με αυτήν και η λογοδοσία σημαίνει ε, σε επίπεδο project, σε επίπεδο δηλαδή έργου, όχι σε επίπεδο χώρας. Οι εκθέσει υποβάλλονται με βάση δηλαδή το έργο. Επίση, έχουμε τι εξαιρέσει από την νομοθεσία τη χώρα υποδοχή. Αυτό είναι κακή ιδέα. Δεν έχουμε στοιχεία ότι η νομοθεσία αυτή θα εμποδίσει τις εταιρείες από το να αποκαλύψουν τις πληροφορίες αυτές. Ε, η Σχολή Νομικής του Κολάμπια, του Πανεπιστημίου Κολάμπια, έκανε μία έρευνα για 150 συμβάσεις και κοίταξε την νομοθεσία σε πολλές ξένες χώρες και δεν βρήκαν στοιχεία ε, νομοθεσιών όπου θα εμποδιζόταν δηλαδή ε, η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν απαγορεύσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας ή επειδή οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικέ, ε, πάντα στις συμβάσεις υπάρχει μια εξαίρεση για τις εταιρείες ε, και οι εταιρείε αυτέ είναι υποχρεωμένε να λογοδοτήσουν Επιτροπή Κεφάλαια Αγορά. Επομένω, να επιτρέψει τι ε, εξαιρέσει αυτέ, επιτρέπει ε, ουσιαστικά στι χώρε αυτέ να αλλάξει νομοθεσία. Και το είδαμε αυτό σε χώρε ακριβώ που μα ενδιέφεραν. είναι κακή ιδέα λοιπόν. Αν θέλουμε τη διαφάνεια να αναγκάσουμε τις χώρες δηλαδή να περάσουν νομοθεσίες τύπου grandfathering. καλό είναι να βάλουμε τουλάχιστον μία προθεσμία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προθεσμία και είναι κακή ιδέα λοιπόν. Ε, θα ήθελα καθώ συζητάτε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που σα είπα να τα λάβετε υπόψη. Αυτά ήταν τα σχολιά μου. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Στίβεν Μπλάιτ από την British Petroleum Company. Τη Βρετανική Εταιρεία Πετρελαίου. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Thank you for this, event. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε να σας ε, παρουσιάσω τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Εξωρετικής Βιομηχανίας. Είμαστε υπέρ της διαφάνειας των δεδομένων και είμαστε πρόθυμοι να αποκαλύψουμε και πληροφορίες για τις πληρωμές και ε, είμαστε υπέρ της εκπόνησης ε, σαφών κανόνων. Να σας πω για το κεφάλαιο 9 πρώτα, για το σχέδιο οδηγίας για τη λογοδοσία. Οι εταιρείε θέλουν να είναι ε, ένα θέμα αναλογικότητας η αποκαλύψη των στοιχείων αυτών για να μην έχουμε ε, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ζημίες ε, εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιριών. Η ε, αποκάλυψη των πληρωμών που αφορούν όλα τα επίπεδα κυβέρνησης θα είναι πολύτιμες πληροφορίες για όλους τους πολίτες και εμείς ε, προτείναμε να υπάρξει μια κατανομή ε, ανάλογα ακριβώς με το επίπεδο διακυβέρνησης, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και επίσης θα πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριε διαγραμμέ του ΟΣΑ. Η πρώτη υποχρέωση των επιχειρήσεων να σέβονται την χώρια νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη απέτηση έχουμε τρει βασικές ανησυχίε. Σε πολλές χώρες οι πληρωμές δεν γίνονται σε επίπεδο έργου, αλλά γίνονται σε επίπεδο συνολικής λειτουργίας μιας εταιρεία στη χώρα. Δεύτερον, ε, δεχτεί και πάρα πολύ δύσκολο να οριστεί ο όρος ε, project, έργο, ε, στις διάφορες χώρες και στις διάφορες εταιρείε. Και τέλος μπορεί να υπάρχει αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών, εταιριών που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη δηλαδή. Και δεν πιστεύω ότι η αναφορά αναέργο είναι ε, βιώσιμη λύση. Τρίτον, η διεύρυνση του κεφαλαίου 9 για να συμπεριλάβει και άλλες χρηματοοικονομικές ε, πληροφορίες, ισολογισμοί, ας πούμε, κέρδη, ζημίες κτλ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι προσπαθώ να καταλάβω ε, πού θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της διαφθοράς η διεύρυνση του κεφαλαίου 9. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω οι πληροφορίες που ζητούνται, πώς βοηθούν και πώς χρησιμεύουν για να καταλάβουν αν πληρώνουν το σωστά ποστά οι εταιρείε. Εγώ έχω διατελέσει και ε, επιθεωρητής ε, και ε, ελεγκτής φορολογικών θεμάτων και σε πολυεθνική εταιρεία και στη δημόσια διοίκηση δεν θεωρώ ότι είναι αυτά τα σωστά μέτρα. Είναι άλλα τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η απαράδεκτη φορολογική ε, συμπεριφορά. Και επίσης η μεθοδολογία πολλαπλής αποκάλυψης. Πολλοί πολιτικοί, υπάλληλοι και εκπρόσωποι εταιριών θεωρούν ότι είναι σημαντικό ε, κάτι τέτοιο να αποφευθεί, να έχουμε κοινά στάνταρ και ε, προδιαγραφές και πρότυπα, Αλλιώ χρειάζεται ε, κάποια συμφωνία αμοιβέ αναγνώριση. Συμπερασματικά θα επανέλθω στο αρχικό μου σχόλιο. Γενικά η εξορρεκτική βιομηχανία είναι υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας. Είμαστε διατεθειμένοι να αποκαλύψουμε τις πληρωμές που έχουμε κάνει προς κυβερνήσεις και με σωστούς κανόνες όμως εφικτούς και εφαρμόσιμους με στόχο η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να γίνει καλύτερη. Ευχαριστώ. Now, Mr. Simon Taylor. Ευχαριστώ κύριο Σάιμον Τέιλερ, Διευθυντής Global Witness που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών. Um, uh, I, want to make... Ευχαριστώ. Τέσσερα σημεία. Θέλω να σας εξηγήσω πόσο καιρό κρατάει αυτή η διαδικασία. Ορισμένοι πρόσφατα ενημερωθήκατε ίσως. Εγώ στο Global Witness ε, ήμουν από εκείνους που ξεκίνησαν ε, την ευστατεία αυτή για τη διαφάνεια το Δεκέμβριο του 1999. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ε, να υποχρεώσουμε την εξορρυκτική βιομηχανία να συντάσσεται σε εκθέσεις. Μιλάμε για 650 μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες προσπαθούν ε, να πετύχουν αυτή τη διαφάνεια. Ε, υπάρχει έλλειψη ε, διαφάνειας για τεράστια κέρδη του εξωρεκτικού κλάδου. Δεν είναι θέμα όμως δεσποτικών ηγετών σε πολλές διεφθαρμένες χώρες, τρίτες χώρες. Υπάρχει και ένα θέμα λογοδοσίας των εταιριών αυτών στο εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να σκεφτούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, διεθνή πρότυπα. Αν τα καταφέρουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, ε, θα κάνουμε απλώς μία φασαρία στο δρόμο, αλλά θα ξεχάσουμε ε, το θέμα της λογοδοσίας των εταιριών. Θα κάνουμε λίγο φτώριβο δηλαδή με διαδηλώσεις και τα λοιπά, τίποτα περαιτέρω. Λοιπόν, θέλουμε να οριστεί σωστά ο όρος project, έργο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, να αναφέρουμε κάποια θέματα, αυτά, αυτά που είπε ο Στίβ, ότι δεν υπάρχει ίδια στάση ε, σε όλο τον κλάδο. Ε, το έργο θα πρέπει να είναι σύνολο δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει δοθεί κρατική άδεια και όπου δίδεται, ε, καταβάλλεται πληρωμή για την άδεια Ε, θα πρέπει να, στις εκθέσεις να αναφέρεται το πώς έχει εξασφαλιστεί η άδεια. Ε, ποια είναι η πληρωμή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Στι αρχέ του 2012, ο θα θυμάται την έκθεση που δημιουργήσαμε για, και που αφορούσε την ε, πληρωμή που δόθηκε από την εταιρεία του στην Αγγόλα. Περίπου 120 εκατομμύρια. Αυτό απαιτείται ε, υποτίθεται δόθηκε για να δημιουργηθεί ένα κέντρο τεχνολογικό, το οποίο όμως δεν δημιουργήθηκε ποτέ, δεν φτιάχθηκε ποτέ. 15 χρόνια χάνει λεφτά η Αγγόλα. Εξαφανίζονται λέει, τα λεφτά. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε έναν ορισμό για το έργο. Ε, εγώ δεν λέω ότι η BP έκανε κάτι παράνομο. Ε, νομικά έπρεπε να το κάνει αυτό. Αλλά μιλάμε για ένα τομέα όπου χρειαζόμαστε μία, μία νομοθεσία πλέον. Στην πρόταση της Επιτροπής υπάρχει μια ρήτρα εξαίρεσης, ε, όπως αυτή που είπε η ε, Διαφωνώ ε, με αυτά που είπε η Σάλη. Ουσιαστικά δίνουμε κίνητρα στους δικτάτορες για να νομοθετούν όπως θέλουν. Ε, νομοθεσίες τύπου Καντάφη κτλ. Ε, τα ίδια κάνει και η Αγγόλα με την ε, Λιβύη. Δεν, ευτυχώς δεν υπάρχει βία στην Αγγόλα, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δικτάτορες που κλέβουν και δεν έχουν καμία, δεν λογοδοτούν πουθενά. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους δικτάτορες να ενεργούν έτσι. Και χαίρομαι που η συγγήτρια, η κυρία Μπράντερ, ε, μίλησε για αυτή τη ρήτρα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξή. Ε, στην έκθεση Λένερ αναφέρθηκε ότι εκεί που οι εταιρείε ε, λειτουργούν σε μια χώρα EITI δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση αποκάλυψης ε, για την πληρωμή. Δεν είναι σωστό αυτό. Πέρα από κάποιες λίγες χώρες σε αυτή τη διαδικασία η e ITI, οι υπόλοιπε δεν δίνουν ε, πολλές προφορίες, οι οποίες είναι απαρχαιωμένες, δεν, είναι, δεν μας λένε τίποτα ουσιαστικά αυτές. Και είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους. Εγώ θέλω να έχουμε στοιχεία ε, καλά, ε, αναέργο, ε, που θα μας λένε κάτι. Και νομίζω ότι με τη σωστά ότι αν δεν του πιέσουμε εμεί αυτού του ανθρώπου, δεν πρόκειται αυτοί οι δικτάτορε οι οποίοι κλέβουν, α πούμε, έτσι από μόνοι του από την καλή του την καρδιά να δώσουν στοιχεία. Επομένω, α του ε, πιέσουμε. last but not least. Ευχαριστώ τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ο κύριο Στέφαν Στέφερ, ο οποίο είναι μέλο συμβούλων σε θέματα management. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ μιλώ ως πρόεδρος του Αφρικανικού Φόρουμ στην ε, ε Βρυξέλλες, που είναι ένα φόρουμ Αφρική. Η διαφθορά είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στις διάφορες αγορές. Θα πρέπει λοιπόν να χαιρετήσουμε την Επιτροπή που έλαβε κάποια βήματα για να μειώσει τις δυνατότητες διαφθοράς δεδομένου ότι υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά πιστεύω ότι οι προτάσεις σε αυτά τα διάγραφα της Κομισιόν είναι ίσως πολύ μετριοπαθή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε, μια θαραλέα, ε, σε ένα θαραλέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επέβαλε διάβια στον τομέα του ανεφοδιασμού σε χημικά προϊόντα. Και δεν μπορεί κάτι τέτοιο προϊόν, εάν δεν έχει ε, υποστεί κάποιες ε, δοκιμασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τεθεί στην αγορά της χημικές βιομηχανίες. Σήμερα, τι βλέπουμε, ότι έχει βελτιωθεί με τον τρόπο αυτό η ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας στην Ευρώπη και ε, με την έβρεση καινοτόμων μεθόδων για την σε, όλη διαδικασία ανεφοδιασμού. Ω κονσάλτα εγώ λοιπόν διαρωτώ με γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε παρεμφερή μέτρα για να μπορέσουμε σε όλες τις αλυσίδες ανεφοδιασμού να μειώσουμε και να καταπολεμήσουμε την ε, διαφθορά. Έχω να κάνω κάποιε. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με την εισηγητρία ότι εδώ θα πρέπει όχι μόνο να συμπεριλάβουμε τον τομέα της εξορρυκτικής βιομηχανία, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί τομείς, οι οποίοι συμμετάσχουν διαφορά στην ε, Αφρική, για να μην αναφέρω τους τομείς των ε, υποδομών, ε, τα θέματα που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα, Πέρσι είχε γίνει μία ε, σχετική έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου για θέματα ειδών διατροφή. Θα πρέπει λοιπόν όντω το θέμα αυτό τη διαφάνεια συμπεριληφθούν όλοι το μίσο Δεύτερον, δεύτερη παρατήρηση. Νομίζω ότι θα πρέπει εκτός από τις ε, κυβερνήσεις, εδώ να συμπεριλάβουμε και όλους τις οργανώσεις και τα κυβερνητικά, δηλαδή ότι οι κλεπτοκράτες δεν είναι ανόητοι, ξέρουν τι ακριβώς συζητείται και στη Washington και στην, ε, ε στις Η κυβέρνηση της ε, ε, Νοτιοαφρικής όλα αυτά τα συμβόλαια και τις ε, συμβάσεις προσπαθεί να τις εξετάσει στα πλαίσια ενός Βουλίου του οποίου ε, ηγούνται κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί το θέμα της ε, υποχρέωσης αναφοράς και η λογοδότηση ξεκινά, η λογοδοσία με συγχωρείτε, ξεκινά από μας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν εμείς τι κάνουμε και γι' αυτό θα ήθελα να υποδείξω το εξής. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να πάρουν το παράδειγμα το οποίο προβλέπει ο Βρετανικός νόμος κατά της δωροδοκίας. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς ενεργούν οι χιλιάδες επιχειρήσεις που καλή την πίστη έχουν το δικό τους μηχανισμό για να αποφευθεί ότι συμμετέχουν σε τέτοιου παράνομες πρακτικές. Ε, υπάρχει και μία ε, στο δικό μας το Αφρικανικό Φόρουμ μια τέτοια πρόνοια, μια τέτοια πρόβλεψη και θα μπορούσατε εσείς να ενθαρρύνετε όλους αυτούς τους μηχανισμούς να τις χρησιμοποιήσουν οι πάντες ώστε να μπορέσουν να ε, δημιουργηθούν θετικά κίνητρα για κάποιον ο οποίος ενεργεί σωστά, διότι οι μεγάλοι επενδυτές όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν ότι υπάρχει μεγάλος πολιτικός κίνδυνος εάν επενδύσουν σε εταιρείε οι οποίες προστρέχουν σε τέτοιου είδους πρακτικές. Πράγμα, αυτό πιστεύω λοιπόν ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτές τις ιδέες. Σας ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι όλοι θα επωφεληθούμε από αυτά ε, τα οποία μας είπατε για να κάνουμε καλύτερη αξιολόγηση του προβλήματος. Η εισηγήτριά μας τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και όλους τους εμπειρογνώμονες. Πολύ ωραία μας περιγράψατε ε, το πλαίσιο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω εγώ και, ε, είναι να σας πω ότι θέλω να υπερασπιστώ στο Κοινοβούλιο. Καλωσορίζω και εγώ πάρα πολύ τις προτάσεις Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής, ακολουθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να μην είμαστε πρωτοπόροι, αλλά ακολουθούμε τους ε, διατλαντικούς μας εταίρους. Και πώς να το πω, για να αποφύγουμε επικαλύψεις και παράλληλες διαδικασίες είναι σωστό και σημαντικό αυτό το βήμα. Ως εισηγήτρια ε, χαιρετίζω λοιπόν και καλωσορίζω πραγματικά αυτή την πρωτοβουλία και είμαι βέβαιη ότι έτσι δεν βοηθούμε μόνο ε, την κοινωνία των πολιτών και τις εταιρείε σε χώρες ε, του τρίτου κόσμου, αλλά βοηθούμε και τους ίδιους μας τους επενδυτές να αποφασίζουν με τα λόγου γνώσεως. Και θα εξασφαλίσουμε και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στον ανεφοδιασμό της ενέργειας, γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα θέματα είναι ε, πιο ασφαλή όταν οι χώρες έχουν ε, κυβερνήσεις που λογοδοτούν και μια σταθερότητα. Λοιπόν, αυτά που κάνουμε για χώρες του τρίτου κόσμου και συγγνώμη που χρησιμοποιώ ε, αυτή την παλιωμοδίτικη έκφραση, αλλά είναι προς αμοιβαίο συμφέρον να προαγάγουμε αυτή τη διαφάνεια στη λογοδοσία. Στην έκθεσή μου εγώ θα επικεντρωθώ βεβαίως σε τρίτες χώρες και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στις τρίτες χώρες. Σίγουρα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη. Δεν πιστεύω ότι θα είμαστε ποτέ σε θέση να εξαλείψουμε πλήρως τη διαφθορά και τη δωροδοκία, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να δυσκολέψουμε τα φαινόμενα αυτά. Γιατί κάποιοι μας λένε ότι δεν θα ξεφορτωθείτε ποτέ, ούτε θα κρυζωθεί η διαφθορά. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δυσκολέψουμε όσο γίνεται τη ε, δυνατότητα ενεργητικής ή παθητικής ροδοροδοκίας. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές σε ορισμένα στοιχεία που ανέφερα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κατόφλι, 100.000 ευρώ για αναφορά πληρωμών. Αυτό νομίζω είναι ένα λογικό επίπεδο και έτσι αποτρέπονται τα βαριά εμπόδια ε, για τα ποσά, ας πούμε, που σε τέτοιους τομείς ε, δεν είναι, σε τέτοιους κλάδους της οικοδομίας δεν πρόκειται για μικρό ποσά. Πάντως, 100.000 μου φαίνεται κατώ, καλό κατόφλι. Επίσης, να ε, απαλληφθεί η ρήτρα εξαιρέσεων για χώρες που έχουν ειδικού νόμους. Δεν χρειάζεται καμία ε, δημοκρατική διαδικασία για να εγκρίνει κάποιο ένα έκτακτο νόμο και γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες στις συμβάσεις τους έχουν ρήτρε που τους επιτρέπουν έτσι και αλλιώ να παρακάμπτουν πολλούς νόμους. Οπότε Και είναι συμφωνία, είναι νόμιμο, γιατί ε, ε, στο συμβόλαιό του το γράφει ότι μπορούν να παρακάπτουν το, το νόμο και έχουν εξαιρέσει, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται αυτό για καμία εταιρεία, από καμία εθνική νομοθεσία. Για μένα είναι σημαντικό αυτό και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνουμε. Άλλο θέμα. Να διευρυνθεί το πεδίο των εταιριών που καλύπτονται και τα δεδομένα που θα πρέπει να αποκαλύπτονται είναι και ο τρόπος εταιρικής διακυβέρνησης μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών που λειτουργούν σε αυτές τις χώρες. Και επίση ε, και εκεί θα πρέπει να ε, μην είμαστε υποκριτές, αλλά συνεκτικοί και συνεπείς στη στάση μας. Και επίσης, αναχώρα, όχι αναέργο, να έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία όπως είναι ο όγκος της ε, παραγωγής και ο αριθμός των εργαζομένων. Όπως είπατε και εσείς, αν έχετε καλύτερες πληροφορίες για το ποιες... Ε, συστάσεις για το ποιες πληροφορίες θα ήταν πιο χρήσιμες να αποκαλύπτονται, δεν έχω αντίρρηση να τα δεχτώ και να βελτιώσω το κείμενο. Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία και είμαι πάρα πολύ υπέρ της προσέγγισης ε, να γίνεται αναφορά με βάση το έργο και όχι τη χώρα. Ελπίζω να με υποστηρίξετε εκεί και ένα τελευταίο για το διοικητικό φόρτο και τα γραφειοκρατικά που θα επιβληθούν ε, στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Το έχω ξανακούσει και σε ιδιωτικές συνομιλίες. Έχω δει πάρα πολλούς ενεχομένους σε αυτή την υπόθεση. Μα δεν χρειάζεται να συλλέγουν νέα στοιχεία οι εταιρείε. Τα έχουν έτσι κι αλλιώς για εσωτερική διαχείριση και για άλλους σκοπούς. Κανονικά κάθε εταιρεία έχει ένα μισολόγιο, ξέρει πόσα χρήματα καταβάλει σε ποιον. Ε, και στο λογιστήριο υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Μπορεί να είναι για εσωτερική χρήση, αλλά δεν χρειάζεται να συλλεγούν εκ νέου. Απλώς να αποκαλύπτονται. και να διαβιβάζονται, γιατί συνήθως αυτά είναι για εσωτερική χρήση και εμπιστευτικά στην εταιρεία. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα γραφειοκρατίας ε, νέας. Και επίσης πιστεύω ότι ακούμε συχνά ότι θα υπάρξουν λέει στρεβλώσεις γιατί υπάρχουν ευαίσθητα στοιχεία και δεδομένα. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, γιατί μίλησα με διαφόρους ε, προσώπους της βιομηχανίας, συνήθως οι ανταγωνιστές ξέρουν σε λεπτομέρειες τι συμβαίνει σε μια εταιρεία. Δεν είναι τεράστιο απόρριτο. Γιατί συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και ξέρουν ε, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές και ε, οι ανταγωνιστές τα γνωρίζουν αυτά εκ Ο έξω κόσμος δεν τα γνωρίζει. Οπότε προσοχή να μην είμαστε ιδιαίτερα <clears throat> υπερβολικά επίοικείς. Και τώρα κάτι προσωπικό. Έχω πάει το τελευταίο εξάμεινο δύο φορές στην ε, Λιβύη και συνάντησα πάρα πολύ θαραλέους νέους που δημιούργησαν ε, τη διαφάνεια της Λιβύης και θέλουν να φέρουν πραγματικά φως σε αυτό το τομέα και έχουν δίκιο. Γιατί αν δεν υπάρχει πουθενά λογοδοσία για το εισόδημα από το πετρέλαιο στη Λιβύη, θα ξαναδούμε την ίδια διεφθαρμένη ελίτ και την ίδια διαδικασία στη χώρα. Και αναλαμβάνουν και πάρα πολύ μεγάλους προσωπικούς κινδύνους. Οι περισσότεροι εργάζονται σε τράπεζες ή σε πετρελοβιομηχανίες και συλλέγουν στοιχεία ε, δικά τους, ε, για λογαριασμό τους και διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο γιατί θέλουν να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια ε, στα θέματα αυτά. Ρισκάρουν τη ζωή τους και θα πρέπει εμείς να δείξουμε ε, παρκές στένος και θάρρος και να τους υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι θα δώσουμε τώρα το λόγο στους συναδέλφους που έχουν γραφεί στη λίστα και μετά σε εσά ε, και στο τέλος στην εισηγήτρια. Ο κ. Πρέντα. Uh, So, around Δύο λεφτά, περίπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητής. Σε σχέση με αυτή την οδηγία για την υποχρέωση αυτή, αλλά εκπροσωπώ τον συνάδελφο, ο οποίος είναι τον κύριο Ουγγουρεάνου, ο οποίο για την δεύτερη οδηγία εισηγητή, που δεν μπορούν να είναι πάρα Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τι δύο γνωμοδοτήσει τη και να ευχαριστήσω και του εμπειρογνώμονες που μα εξέφρασαν τι απόψει του για το θέμα το οποίο μα απασχολεί. Πιστεύω προσωπικά ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τι έχουν να πούν αυτοί οι οποίοι θίγονται άμεσα από αυτές τις προτάσεις και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Στέφεν Μπλάιντ από την BP για την παρουσίαση του. Κατά την άποψή μου, ο εμπορικός τομέας θα πρέπει να εισακουστεί και τα μέλη της Επιτροπής να βρουν μία ισορροπία μεταξύ των πρακτικών θεμάτων που άπτονται αυτών των ε, συμφωνίων διατάξεων και των επιπτώσεων για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και όχι μόνο ε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, και για τους αλλά και για τους υπεργολάβους. Πολλές φορές είναι μικρές επιχειρήσεις. Η ομάδα του ΕΛΚ υποστηρίζει τις εκθέσεις και τη λογοδοσία αναχώρα και έργο Δεν χρειαζόμαστε τριμηνιαίες εκθέσεις. Νομίζω ότι οι εξαμηνίες, οι αιτήσει επαρκούν. Είπα επίσης προηγουμένως ότι το καθεστώς που άπτεται τον ΜΜΕ πρέπει να μας απασχολήσει γιατί αυτές εξαρτώνται από τις μεγάλες επιχειρήσεις και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το θέμα αυτό. Και το ΕΛΚ θεωρεί ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Τώρα, η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο έγγραφο δεδομένου ότι πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ θεωρίας και πρακτικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στις επιχειρήσεις αμερικανικές. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν ε, η οδηγία αυτή και επιχειρήσεις τις οποίες στοχεύει, γι' αυτό θα, στοχεύει, γι αυτό θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ ε, προσεκτικά το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας για να μην ε, πάρουμε αποφάσεις βιαστικές. Ο κύριος Χουίτ, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ κυρία Μπρέτνερ για την εργασία που επιτελέσατε και χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή την κοινή συζήτηση. Κύριε Μπλέικ, Πρέπει να σας συγχαρώ γιατί είστε ο μόνος που δεχθήκατε να μας μιλήσετε υπό την ιδιότητά σας. Θα ήθελα να μου πείτε τι έχει συμβεί με τα 150 εκατομμύρια δολάρια στην Αγγόλα. Εσείς πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ανθίστανται μία επιχείρηση όπως η δική σας δεν θα πρέπει να βλέπει τα πράγματα λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Στην κυρία, αν τώρα θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσει, είπε ο Επίτροπος Μπαρνιέ ότι η Ευρώπη θα ξεπεράσει τους Αμερικανούς σε σχέση με τις απαιτήσει. Τι πιστεύετε εσείς ότι θα γίνει από τη δική σας την άποψη. Όσον αφορά το ρόλο της Επιτροπής, τι μπορείτε να μας πείτε, μπορούμε να βασιστούμε στην εμπειρία των ΙΠΑ. Επίσης θέλω να πω προς όλους ότι εγώ δεν έχω πουθενά οικονομικά συμφέροντα, αλλά μήπως κάνουμε λάθος αν μιλούμε μόνο για την ε, εξορρυκτική βιομηχανία δεν θα πρέπει να μιλήσουμε και για άλλα θέματα και για άλλους τομείς. Τι θα γίνει πίσω κατά την άποψή σας στο Ρίο. Η κυρία Γκόμες για δύο λεπτά. δεν θα εκριζώσουμε τη διαφορά, αλλά μπορούμε να συνεισφέρουμε σοβαρά για την εκριζώση όχι μόνο στι αναπτυσσόμενε χώρε, αλλά και στι δικέ μα χώρε. Δεδομένου ότι η δική του ε, διαφθορά έχει σχέση με τη δική μα και γι' αυτό η έκθεση αυτή είναι τόσο σημαντική και γι' αυτό όντω δεν θα πρέπει κανένα τομέα να τον αποκλείσουμε, καμία χώρα και να μην αποδεχθούμε καμία εξαίρεση στι νομοθεσίε και οι χώρε που έχουν, προβλέπουν τέτοιου εξαιρέσει δεν θα πρέπει να την χάνουν ε, κοινοτικής βοήθειας. Θα πρέπει τέτοιου είδους θέματα να αποτρέψουμε. Και βεβαίως, όντως όπως λέγεται, θα πρέπει για κάθε χώρα να υπάρχει λογοδοσία για κάθε έργο. Θα ήθελα να ότι η χώρα μου, η Πορτογαλία, έχει συγμένες 19 ε, από τις 20 χώρες στο χρηματιστήριο που δεν δημοσιεύουν. Uh, 19 τις 20 εταιρείες που είναι συγμένες στο ε, χρηματιστήριο δεν έχουν τέτοιου είδους ειδικές διαφανείς και λέγουν ότι Βεβαίω υποφέρονται από τα διαφορετικά φορολογικά ευρωπαϊκά συστήματα, από αυτή τη ζούγκλα στην οποία ζούμε, ότι αυτό το κάνουν για να μην ε, δώσουν στην δημοσιότητα ε, όλες τις, ε, τα στοιχεία που αφορούν τις συμβάσεις που τις οποίες κάνουν. Και εδώ αναφέρομαι άμεστο θέμα το οποίο αναφέρθηκε στην Αγκόλα δεδομένες σχέσεις που έχουμε. Υπάρχει λοιπόν στα φορολογικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματική ζούγκλα. Θα πρέπει όμως κάτι να κάνουμε αν θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί με αυτά τα οποία λέμε και για τους άλλους. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτά τα οποία λέγεται για το γραφειοκρατικό άχθος ε, για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη με αφήνει αδιάφορη. Δεν συμμερίζομαι τέτοιου είδους ε, θέματα. Και από την διαφάνεια θα επωφεληθούν όσες επιχειρήσεις ενεργούν με ειλικρίνεια και κυρίως η μιμία. Κυρία Κοπά. Ε, εξετάζουμε σήμερα δύο συναφείς οδηγίες για τη διαφάνεια και την ορθότερη πληροφόρηση και είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση και ενίσχυσή τους στη σημερινή πολύ δύσκολη συγκυρία της οικονομικής κρίσης. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί συνέχεια του έργου που ανελήφθη για την μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και έχει ως κεντρικό στόχο την πρόθεση της διαφάνειας και ψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Και δυστυχώς το θέμα της διαφθοράς παραμένει κεντρικό. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την κυρία Μπραντνερ για την προσέγγιση της πάνω στο θέμα και για τις παρεμβάσεις της στις προτάσεις της Επιτροπής. Οι πληροφορίες πρέπει να διαδίδονται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση για το κοινό και τους μελλοντικούς επενδυτές και εφόσον αυτό είναι δυνατό να φτάνουν οι πληροφορίες τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης αλλά και στο εξωτερικό. Η διασφάλιση της διαφάνειας για τις εξαγορές μεγάλων οικονομικών εταιριών θα συμβάλλει σημαντικά στη χρηματοπιστωτική εξυγίανση και στη σταθερότητα. Η αναγνωρισιμότητα τέτοιου είδους επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο είναι επίσης σημαντική και συμβάλλει ιδιαίτερα στον ανταγωνισμό. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε χώρες όπου δραστηριοποιούνται πολυεθνικές εταιρείες και η διαφάνεια στην υποβολή εκθέσεων χώρα δεν πρέπει να περιορίζεται σε ένα τομέα, ώστε οι επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με την κυρία Μπράντνερ για την ιδέα υποβολής έκθεσης χώρα και όπου απαιτείται και πρόσθετες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον όγκο των εργασιών, αριθμό εργαζομένων κτλ. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εξορρυκτικό κλάδο οφείλουν να δημοσιοποιούν τις πληρωμές που καταβάλουν στις κυβερνήσεις, ανακατηγορία και σε επίπεδο έργου, ως τμήμα της ετήσιας έκθεσής τους. Και είναι σημαντικό οι κανόνες να αφήνουν ένα περιθώριο για περαιτέρω πληροφορίες που μπορούν να ζητηθούν και είναι αναγκαίες για το γενικό συμφέρον ή την προστασία των επενδυτών. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τους κυρίους που παρευρέθησαν εδώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις τους και για μία ακόμα φορά εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να συγχαρώ την εισηγήτρια. Thank you very much. Now, Mr. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Έχετε ένα λεπτό λιγότερο τους άλλους. Ευχαριστώ για τα τρία λεπτά που μου δίνετε. Το πρώτο σημείο. Είναι ένα σημείο που ενδιαφέρει. Πάνω από 200.000 άτομα ζήτησαν τους ηγέτες να λάβουν δράση. Πάνω από 50.000 επιστολές έχουν σταλεί σε ευρωβουλευτές. Ε, όταν σκεφτόμαστε πώς θα βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό είναι ένα θέμα όπου όλοι συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι η διαφάνεια είναι σημαντική. Θα πρέπει να, ε, επίσης να συμφωνήσουμε ότι η νομοθεσία μας είναι σκοπή, ε, υλοποιεί το σκοπό και θα χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Ε, και θέλω να καλύψουμε όχι μόνο βιομηχανίες του εξορρυκτικού κλάδου. Όταν μιλάμε για αυτές, οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες, του εξορρυκτικού κλάδου δηλαδή. Για τον εκπρόσωπο της BP θέλω να του πω ότι έχω μια επιστολή από τον πρώην ε, διευθυντή της BP, τον Λόρδο Τζον Μπράουν. Προφανώς ξέρει πολλά για αυτό το θέμα και άποψή του θα τη διαβάσω, διαβάσω την επιστολή που έστειλε σε έναν υπουργό για αυτό το θέμα. Λέει ότι ορισμένοι από τον κλάδο παραπονούνται ε, για... και θέλουν αδυναμία της, ε, να αποδυναμωθεί μάλλον η πρόταση. Ε, αν δεν θα πρέπει να στα, διασπαστεί ο δεσμός ανάμεσα στο έργο ε, και στον πλούτο που γεννά αυτό το έργο. Ε, επίσης δεν πρέπει να δυσκολευτεί ο τρόπος ε, πληρωμών που κάνουν οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές ε, εισηγμένες εταιρείε. γιατί ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει ένας παγκόσμιος νόμος για την λογοδοσία, κάτι που συζητάει το G20. Με την νομοθεσία αυτή όμως το καταστήσετε αδύνατο αυτό. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ε, υποχρεώσει σε δημοσίευση πριν ε, υπογραφεί το συμβόλιο, η σύμβαση. Το Συμβούλιο προσπαθεί να αποδυναμώσει αυτή την νομοθεσία ε, και κλεισμένων των θυρών θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που θα προκύψει από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο θα είναι να είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ε, και ελπίζω να, καταφέρετε, να το καταφέρετε αυτό. Η κυρία Μπράτνερ έχει ερωτήσεις προς κάποιους από εσά. Θα την υποβάλει, μετά θα απαντήσετε και μετά θα ξαναπάρει το λόγο για τα τελευταία της σχόλια. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Ε, τον εκπρόσωπο της ΒΠ θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί είσαστε κατά της έκθεση έκθεσης αυτής ανά έργο. Ε, για να καταλάβω, γιατί καλύτερα, ποια είναι η αντίρρησή σας που εδράζετε. Ευχαριστώ. Κυρία Χάν. Μετά ο κύριος Μπλάιθ και μετά οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες θα απαντήσουν. Δύο λεπτά ο καθένας. Γρήγορα, λέει η κυρία Χάν θα απαντήσω. Να απαντήσω σε αυτό που είπε η συγκήτρια για την πληρωμή de minimis. Ε, ο γερουσιαστής Καρλέβεν έστειλε στην ε, Επιτροπή Κεφαλαιογράς μια επιστολή για αυτό το θέμα. Είναι πολύ διαφωτιστική και μπορεί να σας δώσει κάποιες πληροφορίες χρήσιμες ε, στις συζητήσεις σας. λέει ότι έγιναν μεμονωμένες πληρωμές, σημαντικές μεμονωμένες πληρωμές, ε, από, λίγα, από χιλιάδες δολάρια ένα μήνα, αλλά οι πληρωμές αυτές αυξάνονται σύν το χρόνο. Ορισμένες είναι, ας πούμε, να πληρώνουν τα δίδακτρα του σχολείου κάποιων παιδιών, ας πούμε, κάποιων αξιωματούχων, ε, φιλοδορήματα, είναι διαφορά δηλαδή. Ε, πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές οι πληρωμές de ε, είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Χάουιτ, ο Επίτροπος Μπαρνιέ στάθηκε στο ύψος της υπόσχεσής του να ξεπεράσει την Αμερικανική νομοθεσία. Ε, γιατί συμπεριλάβει και εμεί συγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείε. Γιατί εμεί περιοριζόμαστε στι συγμένε εταιρείε στο χρηματιστήριο. Μπράβο, μα ξεπεράσατε. Για το ρόλο τη Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά. Είναι σημαντικό να πούμε ότι παρότι καθυστέρησε η εφαρμογή του κανόνα, ε, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι ε, υπήρξε μία δίκη εναντίον της Επιτροπής, ε, γιατί αμφισβητήθηκε το δικαίωμά της να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις. Και αμφισβητείται η οικονομική ανάλυση που γίνεται για τις εταιρείε που είναι η βάση αυτού του νόμου. Έτσι μπλέχτηκε σε αυτό το γκικαιώνα αυτός ο, αυτός ο νόμος, αυτός ο κανόνας. Για το βάρος που θα πέσει στις εταιρείε. Φυσικά, θα πρέπει να δουν οι εταιρείε πώς συλλέγουν τα στοιχεία τους. Θα πρέπει να τα συλλέγουν με νέους τρόπους. Αλλά θα πρέπει, όταν λένε οι εταιρείε όπως η BP ότι θέλουν περισσότερη διαφάνεια, να μας το αποδείξουν τι θέλουν. Ε, και να πούν σε αυτές τις δύσκολες χώρες σε οποίες λειτουργούν αυτές οι εταιρείες όπως η BP, κοιτάξτε, ε, να πούν ας πούμε στους ηγέτες. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε αυτά τα στοιχεία. Αυτό θα πρέπει να τους πούν. Κύριος Μπλάιχ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αρχίσω από αυτό που με ρωτήσατε για τις εταιρείε. Δεν είναι το βασικό επιχείρημα για την Αγγόλα ρωτήσατε που πηγαίνουν τα χρήματα. Είναι υποχρεωμένη η BP ε, βάσει συμβολέου να πληρώσει τη Σόνιγκορ, που είναι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία. Κάθε χρόνο διάφορες ε, πληρωμές γίνονται και στόχος της Sony είναι να τα διαβιβάσει αυτά τα χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι θέμα ε, της BP ε, έχει την υποχρέωση Σόν Αγκόλ να τα δίνει στον κρατικό προϋπολογισμό. Και προτείνεται να αλλάξει η τακτική. Και από ό,τι ξέρω, το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο καταρτίζει μια ενδιάμεση έκθεση ε, και θα είναι αντικείμενο και της έκθεσης αυτής για το αν έχουν χαθεί τα χρήματα αυτά που πήγαν. Δεν έχει λήξει αυτό το θέμα και εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχουν χαθεί χρήματα στην Αγγόλα. Σε ό,τι αφορά την αντίσταση της BP, ε, δεν είναι δίκαιο να λέμε ότι είμαστε κατά των μέτρων. Είμαστε υπέρ ε, της EITI, ε, της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια ε, της εξωτικής βιομηχανίας. Είμαστε σημαντικό μέλος εκεί και σε όλες τις χώρες. Και αν δείτε την ευρωπαϊκή και την αμερικανική νομοθεσία, εμείς συνεισφέραμε ε, με τρόπο ε, επικοδομητικό και σε καμία περίπτωση δεν αντιταχθήκαμε στον νόμο Dodd Frank. Υπάρχουν χώρες που θα γίνουν οι εκθέσεις με τον τρόπο που ισχύει ήδη, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που ε, γίνεται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής ή κρατικής. Και εάν ε, αυτό γίνει αναέργο, ε, θα είναι δυσανάλογη αναφορά ή δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό οι εταιρείε είναι κατά της προσέγγισης της έκθεσης αναέργο και όχι αναχώρα. Αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα υπόλοιποι, παρακαλώ, για δύο λεπτά το πολύ και εσείς. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ. Θα ήθελα οι μεγάλες επιχειρήσεις να είναι, ε, έχουν ίσως διαφορετική μεγίζα από γιατί είναι ίσω ε, λιγότερο διαφορετημένοι. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες που έγιναν σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο οι μεσαίε επιχειρήσεις συμμετέχουν στη διαφορά, Κυρίω εκεί όπου υπάρχει μεγάλη τιμωρησία. Οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις τη χάνουν εποπτείας εκ μέρου των αρχών και οι μεγάλοι επενδυτές της ελέγχους. Και υπάρχουν κανόνες ε, για το πώς ο καθένας ε, ε, επενδύει τα χρήματα. Και ξέρουμε ότι όλο και περισσότερο οι μεγάλες επιχειρήσεις ξέρουν τι επιτρέπεται ή όχι. Πιστεύω όμως ότι συγχρόνως πολλές από αυτές τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ε, και τμήμα στο οποίο ελέγχεται η συμμόρφωση προς τους ε, κανόνες για να ξέρουν πώς θα ενεργήσουν. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο είναι γενικότερο παντού. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία με ισχύ και έξω εδαφική ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν ή να αποτραπούν από τέτοιου είδου πρακτικέ όλε οι επιχειρήσει. Κύριο Τέιλορ, σα ευχαριστώ για την ε, σαφήνεια με την οποία αναφερθήκατε στι πληρωμέ στην Αγγόλα. Αυτό βοηθάει. Αλλά ακούω τι λέγεται εδώ για τις διάφορες ε, πρακτικές και κυρίως αυτή της υποχρέωσης αναφοράς ανά έργο. Θα πρέπει να πω ότι αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε από την άλλη ε, πλευρά του Αντικού εδώ και μερικά χρόνια. Και βεβαίως εκεί τέθηκε καταρχάς ε, θέμα ανταγωνιστικότητας, αλλά είναι και θέμα ε, του ίδιου κανόνα παντού για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πρέπει να πω ότι γενικά οι ε, βιομηχανίες στον ε, πετρελαϊκό τομέα έχουν ε, μία ειδική ε, ίσως νομοθεσία και μεταχείριση σήμερα και σε επίπεδο της ε, American Petroleum υπάρχει τέτοιου είδους ε, πρακτική. Εάν σε κάποιον δεν αρέσει μια νομοθεσία βρίσκει τρόπους να την παρακάψει να την αλλάξει. Το λέγω αυτό διότι αναφέρεται κάποια θέματα τα οποία τα λέτε σωστά. Δεν είναι ε, είσαστε εσείς υπεύθυνοι για την νομοθεσία, αλλά είσαστε υπεύθυνοι για να κάνετε κάτι ώστε να μπορέσει η σωστή νομοθεσία να εφαρμόζεται. ξέρω πώς λειτουργούν οι διάφοροι μηχανισμοί. Όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ίσως δεν ε, καταλαβαίνουμε ε, πώς αντιδρούν, αλλά ξέρουμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά ε, ποσά πολλά εκατομμύρια τα οποία εξαφανίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και γίνονται προσπάθειες τώρα να βρεθούν που πήγανε και με ποιο τρόπο. Διαφορετικά θα έχουμε νομοθεσία η οποία θα έχει εκ πρώτης όψεως τον κατάλληλο χαρακτήρα, αλλά επί της ουσίας δεν θα επιλύει τα προβλήματα. Εάν λοιπόν δεν αρχίσουμε από εδώ να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει, κανένας δεν θα τα κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι καλοί μηχανισμοί, οι οποίοι όχι όμως τύπης, αλλά και επί της ουσίας να επιτρέπουν να γίνεται... Ε, να εμφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Για να ολοκληρώσουμε η Επιτροπή, η κυρία Μπράτνερ. Ο κύριος Κοσμίδης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα λεπτό παρακαλώ. Yes. Ε, Our president, one and a half. Yes. λεπτό. Η κυρία Κοσμίδη, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση εδώ. Ε, ακούσαμε τις διαφορετικές απόψεις εδώ στην ε, αίθουσα. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ πολιτικά φορτισμένο και σκληρό και αυτό προσπαθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξισορροπήσει λίγο την κατάσταση, να προτείνει μια προσέγγιση ισορροπημένη ε, με αναλογικότητα που να φτάνει και στους ε, στόχους μας που είναι να αποθαρρύνεται η δωροδοκία σε τρίτες χώρες και σε χώρες της Ένωσης όμως, όχι μόνο, και να αυξηθεί η λογοδοσία της κυβέρνησης της εκάστοτε. Θα ήθελα να θυμίσω στο κοινό ότι υπάρχει ρήτρα αναθεώρησης στην οδηγία που μπορεί ε, μετά από πενταετία να χρησιμοποιηθεί και ενδεχομένως η πρόταση να επεκταθεί και σε άλλους τομείς μετά από ανάλυση. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να συμφωνήσουμε σε αυτά που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και ουσιαστικά είναι οι τομεί που καλύπτονται από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Τώρα, κυρία Μπράτνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσοι μίλησαν ε, σήμερα και τους εμπειρογνώμονες και ιδιαίτερα από εκείνους που ήρθαν από τόσο μακριά. Και χαίρομαι που ακούω ότι το πρόβλημα δεν είναι το κόστος. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Γιατί κυκλοφορούν πολλές φήμες εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά. Και σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Και προσβλέπω στο κείμενο που αναφέρατε για το κατόφλι ε, έχετε μεγάλη εμπειρία στι Ηνωμένε Πολιτείε και σε τέτοια νομοθεσία και πραγματικά είστε πρωτοπόροι και έχετε ανοίξει τον δρόμο. Ε, βεβαίως οι χώρες ε, είναι δύσκολε χώρε αυτέ που μα απασχολούν. Και ξέρω ότι είναι και πολιτικό πολλέ φορέ το ζήτημα. Οι εταιρείε με την οικονομία ασχολούνται, αλλά σε τέτοιε χώρε δεν μπορούν να αποφύγουν την πολιτική. Και όπως είπε και η Σέλι Χάν, δικό μας καθήκον είναι να δώσουμε αυτή τη ραχοκοκαλιά της ε, νομοθεσίας και να είμαστε στεναροί στην προσέγγιση μας και να δείχνουμε ένα δρόμο προς τα που θέλουμε να κινηθούμε. Το ξέρω, μπορεί ο καθένας να ε, διαφωνεί στον καλύτερο τρόπο της έκθεσης. Στόχος είναι να έχουμε τις πιο καλές προφορίες και τις πιο χρήσιμες προφορίες. Ξέρω και ε, έτσι κι αλλιώς ότι θα γίνουν σκληρές διαπραγματεύσεις και στο εσωτερικό του Συμβουλίου και με το Συμβούλιο. Ε, προσβλέπω στην υποστήριξή σας, τις προτάσεις σας και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ψηφίσουμε. Θα κάνω συνεδριάσει με τους κοιότητες για να καταλήξω σε όσο γίνεται ευρύτερου συμβιβασμός Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ όλους σας για τη συνεισφορά σας. Νομίζω ότι ήταν καλή συζήτηση. Διακόπτουμε τώρα στις 3 και σας ευχαριστώ και τους διερμηνείς.